για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βασιλείου, κύριε Δήμα, στις κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα πολλών συζητήσεων που ήταν και συναισθηματικά φορτισμένες και μπορούμε να ψηφίσουμε δεν φυστήκαμε προσπαθειών και στις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο αναζητήσαμε τις καλύτερες λύσεις. Διαπιστώσαμε ότι η επιστήμη δεν διαθέτει πάντοτε τα πιο ξεκάθαρα διδάγματα. Θα χρειαστεί και άλλη επιστημονική εργασία ώστε να αξιολογηθεί η επίπτωση της νέας αυτής νομοθεσίας. Πρώτα όμως θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν στην προσπάθεια. Τους συναδέλφους μου ευρωβουλευτές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου. Κρίμα που η Τσεχική Προεδρία σήμερα είναι απούσα. Ευχαριστώ και τις συνεργάτες και τους συνεργάτες μας ωστόσο. Κυρίε και κύριοι, με την υποβληθήσα οδηγία για την χρήση των φυτοφαρμάκων κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς περισσότερη ομοιομορφία στο, στην ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας της φύσης για την εξασφάλιση υγιεινών φαρμάκων αλλά και ενός υγιούς περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά η χρήση των φυτοφαρμάκων εναρμονίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική αρχή που λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερα φυτοφάρμακα αλλά να είναι βεβαίως επαρκή γιατί αυτά είναι φάρμακα για τα φυτά και επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο ώστε να αποδίδουν σωστά. Την σωστή χρονική στιγμή πρέπει να δίνεται το σωστό φάρμακο και στην σωστή δόση. Πρέπει βεβαίως να εξετάζεται και το θέμα αν είναι απαραίτητο να ε, γίνει χημική ε, θεραπεία ας πούμε στο φυτό ή αν αρκεί μηχανική και αν εξασφαλίζεται και η καλή εισόδια. Οι χώρες μέλη λαμβάνουν μέτρα στα εθνικά τους σχέδια για την μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ο απότερος στόχος ωστόσο είναι η μείωση του κινδύνου. Από το 2014 θα ισχύσουν οι διατάξεις υποχρεωτικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τήρηση των διατάξεων της Οδηγίας Προστασίας των Ιδάτων έχει πρώτη προτεραιότητα. Η χώρες μέλη ε, δημιουργούν περιθώρια γύρω από τις υδάτινες περιοχές προστασίας τους. Υπάρχουν και διατάξεις για την εξέταση και συντήρηση των μηχανημάτων. Η προσπάθεια που γίνεται για την μείωση του κινδύνου περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των αρμόδιων προσώπων όσοι δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και μπορούν να κάνουν ζημιά χρησιμοποιώντας φυτοφάρμακα έστω και στον κήπο τους, πρέπει ωστόσο να ενημερώνονται από τον πολιτή στο κατάστημα όπου αγοράζουν το προϊόν φυτοφαρμάκου. Με την οδηγία εναρμονίζονται σε ένα υψηλό επίπεδο πολύ διαφορετικές διατάξεις από διάφορες ε, εθνικές νομοθεσίες. Εποφελία του καταναλωτού και του χρήστου. Ίσες διατάξεις εξασφαλίζουν και ίσους όρους ανταγωνισμού. Οι ουσίες εκείνες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι επικίνδυνες πρέπει να απαγορεύονται. Πρέπει ωστόσο αυτά να βασίζονται σε επιστημονικά διδάγματα και όχι σε πολιτικά δόγματα. Το ίδιο σημαντική είναι και η έκθεση των προσώπων στην ε, χρήση των φυτοφαρμάκων. γιατί η δόση βεβαίω είναι αυτή που μπορεί το φάρμακο να το κάνει τελικά δηλητήριο. Έχω έξι λεπτά κυρία Πρόεδρε, έχω έξι λεπτά, έχω και δύο λεπτά από, για την πολιτική, από πολιτική μου ομάδα. Και έρχομαι στο τέλο τη ομιλία μου. Νομίζω ότι ο συμβασμός που επιτύχαμε είναι καλό. γιατί συνδυάζει και την οικονομία και την οικολογία και νομίζω ότι αύριο στην ψηφοφορία θα μπορέσουμε να το τονίσουμε αυτό. Έχω ωστόσο και ένα τεχνικό σχόλιο. Επισημαίνω ένα σφάλμα στο άρθρο 14 παράγραφος 4 όπου γίνεται παραπομπή στην, ε, στο ίντερνετ του άρθρου 4 παράγραφος 3. Όμως το άρθρο 4 δεν διαθέτει παράγραφο 3. Αυτό πρέπει να διορθωθεί λοιπόν εξ αρχής. 5 λεπτά κυρία Κλάς θα διερευνήσω να δω αν έχετε περιθώριο να παρέμβετε και στο τέλος. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπρέγερ, παρακαλώ. Για τέσσερα λεπτά, κυρία Μπρέγερ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ε, κυρία Επίτροπε, αγαπητή κύριε Επίτροπε, η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για την προστασία της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την οικονομία. Πρώτα, ευχαριστώ ιδιαίτερα την σκιώδη συγκήτρια και τον σκιώδη συγκητή για την εξαιρετική συνεργασία που μου προσέφεραν. Ευχαριστώ βεβαίως και όλα τα πρόσωπα που συνεργάστηκαν ε, για την σύνταξη του κειμένου. Και βεβαίως ευχαριστώ και ιδιαίτερα εσάς, κυρία Βασιλείου, και εσάς, κύριε Δήμα, αλλά και την Γαλλική Προεδρία. Επίσης, ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους εκείνους που ε, δεν ε, πανικοβλήθηκαν από την ε, πίεση λόμπι της βιομηχανίας. Στην πρώτη ανάγνωση είχαμε 200 τροπολογίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ψηφίσαμε σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου. Με ξεκάθαρα κριτήρια cut-off που σταματήσαμε τον τρόπο αυτό όλα τα αμπρακατάμπρα και τα χόκους πόκους της βιομηχανίας. Κανείς δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει τον κίνδυνο. Γι' αυτό είναι καλύτερα να υπάρξει μια πλήρης απαγόρευση. Καρκινογόνες, ουσίες στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχουν απολύτως κανένα ρόλο να παίξουν μέσα στα φάρμακα. Με αυτό το κάτω για τα PPT φροντίζουμε ώστε να είναι επιτυχής η προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα με χαροποιεί το γεγονός ότι μπορέσαμε για πρώτη φορά να θεσπίσουμε σαφή κριτήρια για ε, ε, ουσίες οι οποίες επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου. Και ελπίζω ότι θα μπορέσει αυτά να τα περιλάβει και στις μελλοντικέ προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα με ικανοποιεί επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτυχε για πρώτη φορά και πάλι την προστασία των μελισσών να την βάλει ως σαφές κριτήριο. Υπάρχουν επιστήμονες και στην Γερμανία και στη Γαλλία που ε, αξιολογούν τις σχετικές ζημίες σε 150 δισεκατομμύρια τον χρόνο και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημία εάν οι ε, μέλισσες δεν μπορούν πλέον να παίξουν τον ρόλο της γονιμοποίησης των φυτών με τη γύρι. Υπάρχουν ορισμένοι που προσπαθούν να αποδυναμώσουν τον συμβιβασμό. Όμως εγώ επισημαίνω ότι το Συμβούλιο ήδη έχει δεχθεί τον συμβιβασμό αυτό και δεν θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ανατραπεί. Χαίρομαι πάντως και για το γεγονός ότι με κοινή προσπάθεια μπορέσαμε να επιτύχουμε και μια βελτίωση για το θέμα των ανοσοτοξικών ουσιών. Γιατί σε μια Ευρώπη που θέλει να είναι κοινωνία της γνώσης δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτές οι ανοσοτοξικές ουσίες να κάνουν ζημιά στην εξέλιξη του εγκεφάλου των παιδιών και μάλιστα με τρόπο βαρύ και διαρκή. Λέμε λοιπόν ναι στην εναρμόνιση χωρίς ωστόσο να περιορίζουμε το δικαίωμα των χωρών μελών σχετικά με την έγκριση κυκλοφορίας των ε, προστατευτικών προϊόντων. Δείχνουμε με τον τρόπο αυτό τι μεγάλη αξία αποδίδουμε στην υγεία. Έχουμε, και δυνατό, έχουμε προβλέψει και δυνατότητα υποκατάστασης ώστε να μην γίνει η εξαίρεση ο, κανόνες, ο κανόνας. Και χαίρομαι επίσης που μπορέσαμε να περιλάβουμε στον κανονισμό αυτό και την προστασία των ζώων και ότι εξασφαλίσαμε περισσότερη διαφάνεια. Παρόλο που εγώ θα είχα προτιμήσει να είχε δείξει περισσότερο θάρρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω πάντως με αυτή την μεγαλύτερη πρόσβαση στα πρωτόκολλα χρήσεως να ε, μπορέσουμε να το επιτύχουμε να μπει και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, η τελευταία φράση που έχω να πω είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για ορόσημο για το περιβάλλον και την προστασία του καταναλωτού στην Ευρώπη, πρόκειται πραγματικά και για μια κορυφαία στιγμή της Ευρώπης. Κορυφαία λέγω διότι αυτή η απόφαση να αποκλειστούν τα βαριά αυτά και επικίνδυνα φυτοπροστατευτικά φάρμακα είναι πρωτοφανής στον κόσμο και οδηγεί σε πρωτοπορία την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολόκληρο τον κόσμο και νομίζω ότι δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία υπέρ των πολιτών που γνωρίζουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπαραταχθεί μαζί τους με τους καταναλωτές, με τους πολίτες και βάζει φραγμό στις προσπάθειες της βιομηχανίας που άλλωστε είναι αμοιβαία υποφελής και για τη βιομηχανία η οποία στο μέλλον θα μπορεί να παράγει πιο ασφαλή προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι για τον χρόνο ομιλίας των εισηγητριών. Ε, μιλήσατε πέντε λεπτά, η κυρία Κλάς έχει άλλο ένα λεπτό το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο τέλος, δεν έχει χρόνο από την πολιτική ομάδα και η κυρία Μπρέγκερ έχει, μίλησε 5,5 λεπτά, έχει 1,5 λεπτό στην πολιτική ομάδα και τα δύο λεπτά στο τέλος. Τώρα ο κύριος Δήμας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια κυρία Βασιλείου. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Κλάς την εισηγήτρια κυρία Μπρέγερ, καθώς και την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου για την εξαίρετη εργασία τους σχετικά με τις ε, προτάσεις αφενός για την οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων αλλά και για την αναθεώρηση και βελτίωση του κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει την περιβαλλοντική ακεραιότητα της αρχικής πρότασης της επιτροπής ενώ σε ορισμένα σημαντικά σημεία θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους. είναι γνωστό ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους πολίτες. για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητο αφενός μεν να καταστεί αυστηρότερο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με την τροποποίηση της οδηγίας του 1991 για τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά αφετέρου δε να συμπληρωθούν τα κενά που παρατηρούνται σε κοινοτικό επίπεδο κατά το στάδιο της χρήσης των εν λόγω προϊόντων. με την επίτευξη συμφωνίας για την οδηγία η ευρωπαϊκή ένωση αποδεικνύει ότι έχει την πολιτική βούληση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος το κοινοβούλιο συνέβαλε ώστε η οδηγία σε ορισμένα σημαντικά σημεία να είναι πιο φιλόδοξη από την κοινή θέση του συμβουλίου. πιο συγκεκριμένα τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταρτήσουν εθνικά σχέδια δράσης με ποσοτικούς στόχους τόσο για τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει η χρήση φυτοφαρμάκων όσο και για την μείωση της χρήσης ορισμένων προϊόντων. αυτό δεν ήταν εύκολο ε, καθώς η εισηγήτρια έπρεπε να πείσει τα κράτη μέλη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ενδεδειγμένο ε, μέσο περιορισμού του κινδύνου είναι η μείωση της χρήσης συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων. αυτό το έπραξε με επιτυχία. η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί σημαντική πρόοδο για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος στην ευρωπαϊκή ένωση. συνεπώς η ευρωπαϊκή επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη τροπολογιών ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την οδηγία σε δεύτερη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Βασιλείου. Το κυρία Πρόεδρε. members. Καταρχήν, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες, της κυρίας Κλάς και Μπράγερ και του Σκιώδης για την επικοδομητική του προσέγγιση στην πρόταση όπως και τη Γαλλική Προεδρία και όλους εσάς που συνεισφέρατε στην επιτυχή διεκπαιρέωση της δεύτερης ανάγνωσης της πρότασης Επιτροπής. Όπως ξέρετε, τα προϊόντα, τα φυτικά αυτά προϊόντα παίζουν σημαντικό ρόλο και στην κυπευτική και στην γεωργία και στη δασοκομεία, αλλά μπορούν να έχουν επιπτώσεις και στη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό θα πρέπει να διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς που να εξορροπεί την κατάσταση. Κατά την ε, προετοιμασία της αρχικής πρότασης είχαμε μακρές διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και προωθήσαμε μία εκτενή μελέτη αντικτύπου. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος. Χαίρομαι διότι αυτό αντικατοπτρίζεται και από τη συζήτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων και θεσμικών οργάνων. Η πρόταση αυτή συμβιβασμού θα ενισχύσει αυτή την προστασία με συγκεκριμένες διατάξεις. Θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για την έγκριση των ενεργών ουσιών Επίσης, οι παραγωγοί, οι προμηθευτές και οι επαγγελματικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν μητρώα τα οποία θα μπορούν να διαθέσουν σε τρίτους, σε περίκους και σε μέλη διαφόρων οργανώσεων που ασχολούνται και με τον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης, θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνονται, έτσι δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις και διασταυρούμενες έρευνες. Επίσης θα έχουμε ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για τα πιο επικίνδυνα προϊόντα. Για να υπάρχει εκτενής πληροφόρηση, η Επιτροπή θα ασχοληθεί και με την διαθεσιμότητα εναλλακτικών προϊόντων σε σχέση με ουσίες που θεωρούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες. Αυτό θα γίνει χωρίς να προδικάσουμε τις προδιαγραφές ασφάλειας του κανονισμού. Στα πλαίσια του ολικού συμβιβασμού θα ήθελα να προτείνω το εξής κείμενο σε σχέση με την ε, εκτίμηση κινδύνου όταν αναθεωρούνται τα στοιχεία για τις ενεργές ουσίες και τις, ε, τα προϊόντα όπως αναφέρονται στις παραγράφους 8α και γ, η Επιτροπή θα προσδώσει μεγάλη σημασία στη μελέτη πρωτοκόλων έτσι ώστε να γίνει επανεκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική έκθεση σε αυτά τα προϊόντα, ιδιαίτερα ε, μέσα από την γύρι και το νέκταρ. Επίσης, θα υπάρχει ένα σαφέστερο πλαίσιο για την προστασία αυτών των, προϊόντων στην, ε, των φυτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής προστασία και του περιβάλλοντος και των πολιτών. Επίσης, θα αντικατοπτρίζεται η στρατηγία της Λισαβόνας μειώνοντας τη γραφειοκρατία έτσι ώστε η διαδικασία να είναι βραχύτερη και πιο αποτελεσματική η διαδικασία έγκρισης. Επίσης τα κράτη-μέλη δεν θα εργάζονται ε, απομονωμένα το ένα από το άλλο, διότι θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Επίσης δεν θα υπάρχει κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς και θα υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα παρασιτοκτόνων για τους αγρότες. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία ε, οδηγία για την ε, αηφόρο χρήση των ε, παρασιτοκτόνων που εμπίπτει στη δραστηριότητα του κυρίου Δήμα. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η κυρία Χένικοτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους και τον Επίτροπο και την Επίτροπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις εισηγήτριες και ιδιαίτερα την Γαλλική Προεδρία η οποία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να εξευρεθεί αυτή η συμφωνία, ο συμβασμός που βοηθά στην ανθρώπινη υγεία. Μιλάμε για ένα τριζωνικό σύστημα το οποίο θα βελτιώσει την προσπελασιμότητα στα προϊόντα και επίσης ε, ε, μιλάμε και για την ε, χρήση προϊόντων για, για ελάσσονες καλλιέργειες και για προϊόντα κυπευτικής. Μιλάμε επίσης για την προθεσμία του 2020 για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα CMR. Έτσι θα μειωθούν οι ασθένειες και οι νεοπλασίες που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα κάτι το οποίο έχει ε, αποδεκτεί επιστημονικά. Και αυτό αφορά και άλλες μορφές ασθενειών. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας και για την ε, μελισσοκομεία. Η Επιτροπή έχει προβεί σε μία δήλωση επί του θέματος και θα ήθελα να μου πει κατά πώς θα λάβει υπόψη την οδηγία 2007 κάθετος 52. Επίσης θα τονίσουμε τις ε, διάφορες ε, μορφές ε, θέσεις εμπορία προϊόντων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή. Έτσι, θα προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία ως προς τις ε, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα παρασιτοκτόνα. Θα υπάρχουν και ενδιάμεση έλεγχοι και ελπίζω ότι οι εθνικές αρχές θα μπορέσουν να αποδείξουν την αξιοπιστία του κειμένου. Σοσιαλιστικής ομάδας, ο κύριος Γόργενσεν, για ε, τρία λεπτά. ευχαριστώ, for formand. Da forslaget fra kommissionen blev offentliggjort, der όπως ξέρετε, η πρόταση της Επιτροπής ε, δημοσιεύτηκε ήδη και ε, οδήγησε σε συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τον υδροφόρο ορίζοντα και αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση ερχόμαστε σε έχουμε άμεση σχέση με τον υδροφόρο ορίζοντα και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει πληγεί από τα διάφορα φυτοφάρμακα. Πολλά φυτοφάρμακα φιλτράρονται στον ε, υδροφόρο ορίζοντα, άρα το νερό αυτό δεν είναι πλέον πόσιμο. Αυτό ακριβώς μας απασχολεί και αυτή ήταν και η αρχική πρόταση της, και της Δανίας και της Επίτροπης. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς που θα πρέπει να τύχουν της προστασίας μας. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθησε για να φτάσουμε σε αυτό το ευέλικτο πλαίσιο έτσι ώστε κάθε χώρα να μπορεί να απαγορεύσει ένα φυτοφάρμακο που την χρήση του οποίου δεν επιθυμεί. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι και η απαγόρευση των ε, πιο επικίνδυνων ίχνοστοιχείων ενός φυτοφαρμάκου. Αυτό γίνεται και μέσα στα πλαίσια του REACH. Άρα δεν θα επιτρέψουμε μία σειρά ουσιών στα παιχνίδια ή στα είδη ένδυσης, αλλά μπορούσαν να ενυπάρχουν στα φυτοφάρμακα. Έτσι μπορούμε να άρουμε αυτό το πλαίσιο χρήσης ε, στα φυτοφάρμακα και αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν και τα εθνικά σχέδια ή προγράμματα όταν μιλάμε για συστήματα μέτρησης επικινδύνων ουσιών στα φυτοφάρμακα. Υπάρχουν ουσίες που είναι πλέον επικίνδυνες από άλλες και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ποσοτική χρήση των φυτοφαρμάκων που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Νομίζω λοιπόν ότι το έγγραφο είναι πολύ καλύτερο και τα νεοτοξικά αυτά προϊόντα θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα για την προστασία των παιδιών, ως προς την προστασία των παιδιών. Επίσης, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος ως προς τις εξαιρέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιτελεστεί μεγαλύτερη πρόοδος. των κυρία για τέσσερα Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στη... στο σημείο έγκρισης αυτών των δύο εκθέσεων για τη χρήση φυτοφαρμάκων. Νομίζω ότι πρόκειται για μια εξορροπημένη προσπάθεια που θα πρέπει να υποστηριχθεί. Για τους παραγωγούς και τους χρήστες έχουν γίνει πολλές πρόοδοι. Μιλάμε για την απλούστευση της, ε, του γραφειοκρατικού πλαισίου και της διοικητικής έγκρισης με βάση ένα τριζωνικό. Θα ήθελα να είναι μονοζωνικό όμως το σύστημα, αλλά τα κράτη-μέλη ε, δυστυχώς δεν το δέχτηκαν. Ήταν επιφυλακτικά. Αυτό αφορά και τους πολιτές και τους χρήστες. Θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα φυτοφάρμακα και αυτό και για οικονομικούς λόγους. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προστασία όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των ζώων. Και αυτό το είδαμε μετά από δοκιμασίες που έγιναν. Μας ενδιαφέρει και η προστασία του περιβάλλοντος βεβαίως γιατί οι πιο επικίνδυνες ουσίες θα αντικατασταθούν από λιγότερο επικίνδυνες. Επίσης υπάρχει και το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα νομικό κείμενο που να ασχολείται με αυτό τον ορισμό. Η Επιτροπή έχει τέσσερα χρόνια για να υποβάλει προτάσεις μέτρων με επιστημονικά δεδομένα για να ορίσουμε αυτές τις ιδιότητες που ορίζουν του, τις ενδοκρινικές διαταραχές. Έτσι ώστε, de facto, η φάρμακοβιομηχανία να έχει και ένα νομικό πλαίσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις μέλισσες και τον ρόλο του στο οικοσύστημα. Φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό με βάση αυτό το επιπρόσθετο κείμενο. Πιστεύω ότι οι ενεργές ουσίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτό αφορά ιδιαίτερα τη γύρι και τον νέκταρ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ενεργές ουσίες και πολλοί ε, αναφέρθηκαν σε αυτές. Πιστεύω ότι το τριζωνικό σύστημα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερα προϊόντα και υπάρχει και δυνατότητα εξαίρεσης σε σχέση με τις ελάσσονες χρήσεις θεωρήσαμε ότι βράχει πρόθεσμα η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις και ως προς ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο υπάρχει και η ρήτρα επανεξέτασης έτσι ώστε η Επιτροπή να δει κατά πόσο υπάρχει σωστή διαφοροποίηση και ανταγωνισμός της γεωργίας. Τέλος, και αυτό υπενθύμησαν οι συνάδελφοι, θα θέλαμε οι παρασκευαστές φυτοφαρμάκων να προωθήσουν νέα προϊόντα που να σέβονται την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, τα προϊόντα αυτά, τα φυτοφαρμακευτικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, με σωστή και λογική χρήση και πιστεύω ότι έτσι θα υπάρχει ολοκληρωμένη χρήση για μία αηφόρο γεωργική ανάπτυξη. Έτσι θα φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση ως προς την προστασία της υγείας και την διαθεσιμότητα προϊόντων για τους αγρότες. Αγαπητοί συνάδελφοι, χάρηκα ιδιαίτερα που μπορέσαμε να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να έχουμε μια σωστή επαφή και θα ήθελα να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες, Κλάς και Μπράγερ, οι οποίες ήταν πολύ σωστές διαπραγματεύτριες κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Το λόγο τώρα θα πάρει ε, για τρία λεπτά εκ μέρους της Ένωσης για την Ευρώπη των Εθνών ο κύριος Άιλουαρντ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλούμε παραμονές σημαντικής ψηφοφορίας για τη Γεωργία, για την Υγεία και το περιβάλλον να είναι ξεκάθαρο κάτι. Οποιοδήποτε από εμά του νομοθέτε που έχει εντοπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια τη νομοθετική διαδικασία το έκανε αυτό διότι ανησυχεί για τη γεωργία και για τη μελλοντική παραγωγή τροφίμων. Βεβαίω ανησυχώ για οπουδήποτε υπερβολική χρήση των παρασυντοκτώνων και των συνεπειών του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα καρκίνων. Έχουμε αυξήσει τα κατάλοιπα στα τρόφιμα, στον αέρα και στο νερό. Και αυτό επηρεάζει τη υγεία και το περιβάλλον. Και η γεωργοί μα είναι σε καθημερινή επαφή με τα βασιτοκτόνα και επηρεάζεται περισσότερο. Λοιπόν, η νομοθεσία θέλει να προστατεύσει την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον και τη γεωργία. Σαν νομοθέτε όμω θα πρέπει πάντα να πετυχαίνουμε ισορροπία και να βασίζουμε σε επιστημονικά στοιχεία την νομοθεσία μα. Δεν μπορούμε και θα πρέπει να νομοθετούμε έτσι αφηρημένα συγκεκριμένα Αποκρινόμενοι από την αρχική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλυση του κινδύνου, ε, τελικά πέσαμε στο πρώτο εμπόδιο. Χωρίς αξιολόγηση του κινδύνου που πολλοί από εμάς ζητήσαμε επανειλημμένα, κανείς δεν μπορεί να δηλώσει επακριβώς πόσες ουσίες θα απαγορευτούν. Η Ιρλανδία έχει ένα ήπιο κλίμα, υγρό, Οπότε τα δημητριακά, τα χειμωνιάτικα και οι πατάτες ε, έχουν διάφορα προβλήματα από διάφορα παράσιτα. Εάν βγάλουμε λοιπόν διάφορα προϊόντα που δεν θα έπρεπε, θα επηρεαστεί η παραγωγή των προϊόντων. Σε 18 μήνε θα, εισαχθεί, θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Τι θα γίνει, τα παρασιτοκτόνα που με την παρούσα νομοθεσία επιτρέπονται θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι να εκπνεύσει η αδειοδότησή τους. Αν στην Ιρλανδία μπορούμε να αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη ουσία που θα πρέπει να αποσυρθεί χρειάζεται για την καταπολέμηση σοβαρή ασθένεια των φυτών, και δεν υπάρχει υποκατάστατο ασφαλέ. αυτή η ουσία μπορεί να εγκριθεί επανειλημμένα για μια πενταετία παρά την απαγόρευση. Θεωρητικά αυτό μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, θα πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει. Με το παρόν κλίμα δεν μπορούμε να μειώσουμε την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά. Θα πρέπει να προωθήσουμε τον τομέα γεωργία να παράγει προϊόντα και να χρησιμοποιεί εναλλακτικά προϊόντα που θα είναι εξίσου αποτελεσματικά, αν όχι περισσότερο. Είδαμε τι έγινε όταν χρησιμοποίησαμε διάφορα φάρμακα ε, που ήταν ε, για να προστατεύσουμε τα άσπρα στα φύλλα. Μέσω των τροπολογιών μας μπορούμε να προστατεύσουμε την επικονίαση μέσω των μελισσών. Θα ήθελα να υποστηρίξετε την τροπολογία 182 και να αποσυθεί η 169. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπειρογνώμονες θα δώσουν τη σωστή επιστημονική βάση ούτως για τους ενδοκρινικούς διαταράχτες με τετραετία. Δεν θα μπορούσαμε να προδικάσουμε επιστημονικά πορίσματα με ενσωμή επιστημονικού ορισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για την ομάδα των Πρασίνων η κυρία Μπρέγερ, για δύο λεπτά. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω για την έκθεση της κυρίας Κλάς, αλλά με την ευκαιρία θα απαντήσω στον συνάδελφό μου που μίλησε πριν παρακαλώ διαβάστε την συμφωνία. Εμείς καταθέσαμε την τροπολογία ώστε οι ε, ε, ουσίες που θίγουν το ενδοκρινικό σύστημα να μην μείνουν άλλα τέσσερα χρόνια. Αυτό όμως επιδιώκει η τροπολογία σας. Επειδή λοιπόν είναι αντιφατικό με αυτό που είπατε, παρακαλώ την επανεξετάσετε. Και βέβαια Άλλη υπόθεση, εάν θα υποκληθούμε στην ε, βιομηχανία που παράγει φυτοφάρμακα ή εάν θα ε, ορθώσουμε το παράστημά μας για να προστατεύσουμε τους πολίτες και τους καταναλωτές. Και το παράδειγμα που ανέφερε προηγούμενα άλλος συνάδελφος, όπου μέσα σε 20 χρόνια μπόρεσαν να μειώσουν κατά το ίμιση την χρήση ε, φυτοφαρμάκων και να βελτιώσουν την ε, ποιότητα των υδάτων. Για λίγα δευτερόλεπτα να μιλήσω για την έκθεση της κυρίας Κλάς. Αφού την ευχαριστήσω πρώτα για την εργασία της, θα θέλαμε βέβαια, όπως είπα, να είχαμε ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε ότι ε, η έκθεσή σας, η οδηγία, θα αποτελέσει προτροπή και για τις ε, χώρες μέλη να ακολουθήσουν αυτές τις άλλες χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν περισσότερο. Και βέβαια θα θέλαμε να υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα για τους κατοίκους ε, περιοχών γειτονικών με ε, γεωργικές περιοχές και υπενθυμίζω και την απόφαση του Ανώτατου Βρετανικού Δικαστηρίου που υποστηρίζει τους πολίτες στην αξίωση που προβάλλουν να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες μπορούμε να βασιστούμε στην απόφαση αυτή ώστε να κάνουμε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε περισσότερη πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ελπίζω μάλιστα να οδηγήσει αυτό και σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ κυρία Μπρέγκερ. Ο κύριος Μουσάτσιο από την ε, Ενωμένη Αριστερά για δυόμιση λεπτά. Ε, η αντιπαράθεση από αυτών διατάξεων για την παρασιτοκτόνο υπήρξε πάρα πολύ σκληρή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε σωστά για νομοθεσία που θα πρέπει να φασιστική και να καλύπτει τα προβλήματα. Ακολουθήθηκε διαλεκτική κοινοβουλευτική, αλλά κυρίω υπήρξε ισχυρή αντίσταση στο Συμβούλιο. Και υπήρξαν οικονομικά συμφέροντα που κινητοποιήθηκαν για να προστατευτούν θα πρέπει αντίθετα να εξετάσουμε τα γενικά συμφέροντα. Αυτό το καταναλωτών που θέλουν να τρώνε τρόφιμα που δεν είναι μολυσμένα. Οι πολίτε που θέλουν ένα περιβάλλον που δεν πλήττεται από αυτά τα παρασιτοκτόνα. Του γεωργού που θέλουν να εργάζονται ασφαλώ και θα θέλουν να έχουν νέα ποιότητα στα προϊόντα του. Υπάρχει υπερβολική χρήση χημικών ουσιών στην γεωργία που βλέπει του πάντε. Το τρόφιμα, το περιβάλλον, του γεωργού που θα πρέπει να πληρώνουν ακριβά αυτά τα βιομηχανικά προϊόντα. Λοιπόν, είναι παλιό το μοντέλο η χρήση των χημικών. Δηλαδή είναι η γεωργία της ποσότητας και της ποιότητας. Τα προϊόντα διαχωρίζονται από την ύπεθρο, από τις εποχές και από τη δουλειά. Δαπανηρό μοντέλο για όλους. Ευλαβές, ε, διότι επηρεάζει και δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτή η νομοθεσία εντάσσεται στη δημιουργία υγιέστερου και πιο σύγχρονου μοντέλου. Μια γεωργία ποιοτική θέλουμε, όπου οι πολίτες και το περιβάλλον προστατεύονται και έχουμε θέσει εργασία στη δουλειά που κάναμε πετύχαμε θετικά αποτελέσματα. Χάρη στην επιμονή και των δύο συγγετριών και όλου του τεχνικού προσωπικού που, αντιμε... που ήρθε σε επαφή με τους συναδέλφους τους του Συμβουλίου. Ο στόχος της μειώσεως της παρουσίας παρσιτοκτόνων και όχι μόνο λόγω επικινδυνονότητας εισήχθη μόνο διότι θέλαμε να κινηθούμε σε εθνικά πλάνα, κυρίως όσον αφορά τις ουσίες ψηλού κινδύνου. Λοιπόν, θέλουμε μη χημικές μεθόδους για την προάσπιση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα και θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το κοινό αγαθό το νερό. Άρα θα πρέπει οι διάφορες χώρες να καταλάβουν ποια μεγάλη ευθύνη υπέχουν όσον αφορά τη χρήση των παρασιτοκτόνων. Λοιπόν, απαγορεύεται ο ψεκασμός από τον αέρα. Και θα πρέπει λοιπόν, εάν γίνει ο ψεκασμός, να ενημερώνεται δεόντως έγκαιρα ο πληθυσμός έγιναν ε, πρόοδοι όσον αφορά την ενημέρωση και στην πρόσβαση στα στοιχεία μέσω του διαδικτύου. Θέλαμε έναν κανονισμό όπου εγκαταλείπτεται η ιδέα των τριών ζωνών. Όμω λόγω Συμβουλίου παρέμεινε αυτό ο διαχωρισμό. Τα αποτελέσματα όμω είναι σημαντικά. Τα μέτρα αυτά θα εθετηθούν για την καταπολέμηση τη παράνομη χρήσεω των επικίνδυνων ουσιών. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό βήμα πρόοδου και ελπίζω ότι η ψηφοφορία δεν θα οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες. Ο κύριος Μπλόκλαντ από την ομάδα Ανεξαρτησία Δημοκρατία για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση όσον αφορά τη διάθεση των φυτογενομικών προϊόντων είναι δύσκολη συζήτηση, δύσκολη ισορροπία μεταξύ καλών και κακών στοιχείων. Οι χημικές ουσίες βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον. Η γεωργία όμως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς παρασιτοκτόνα διότι θα είχαμε προβλήματα ίσως για την υγεία των φυτών. Και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων και όσον αφορά την οικονομία. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας από τη μία και της γεωρικής οικονομίας από την άλλη. Αυτή η συμβαστική πρόταση ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση ισορροπίας. Γι' αυτό την ε, υποστηρίζω. Χαίρομαι που ε, μπορέσαμε να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που οδηγεί στη μείωση του κινδύνου και όχι τη μείωση της χρήσης. Η μείωση της χρήσης δεν συνεπάγεται αυτόματα και την μείωση ε, του κινδύνου αν μειωθεί η ποσότητα των ουσιών, αλλά χρησιμοποιούμε τις ουσίες αυτές σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, αυτό δεν κάνει και πολύ μεγάλο καλό στο περιβάλλον. Χαίρομαι που ο κανονισμός όσον αφορά την αδειοδότηση δεν είναι τόσο περιοριστικός όπως στην πρώτη ανάγνωση. Επιβάλλονται ε, νέα όρια όσον αφορά την αδειοδότηση των ουσιών, αλλά αυτό δεν θα επιφέρει σημαντικές ζημίες στην Γεωργία. Ευχαριστώ τους συζητητές για τη συνεργασία και τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Ευχαριστώ. Τώρα από τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Μόουτ για 1,5 λεπτό. I have been deluged Έχω κατακλειστεί από μηνύματα από διάφορους ε, παραγωγούς και καλλιεργητές που θεωρούν αυτή την ε, πρόταση ε, άκρος καταστροφική. Γιατί θα έχουμε μικρότερες καλλιέργειες, υψηλότερες τιμές και έτσι οι εισαγωγείς που δεν ακολουθούν τα ίδια κριτήρια θα μπορούν να κατακλείσουν την αγορά, θα χαθούν, θα χαθούν θέσεις εργασίας πολλές, πολλές παραγωγές θα σταματήσουν, θα κλείσουν εργοστάσια στη δική μου εκλογική περιφέρεια, διότι σε ορισμένες ε, περιπτώσεις δεν υπάρχουν εναλλακτικέ σε σχέση με τις ενεργές ουσίες που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί. Δυστυχώς ε, δεν έγιναν σωστές μελέτες αντικτύπου σε πολλές χώρες, εκτός από τη δική μου, και μιλάμε και για την αποτίμηση κινδύνου. Εάν χρησιμοποιήσουμε τον κίνδυνο ως ε, κριτήριο, τότε ας απαγορεύσουμε και την καφέινη και το πετρέλαιο. Ακόμα και η επιστήμη σας αντιτάσσεται, διότι ξέρετε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα ζυζάνια. Δεν θα υπάρχει βιοπικιλότητα πλέον και επίσης τα ολοκληρωμένα προγράμματα ε, ανάπτυξης φυτών δείχνουν ότι δεν χρειάζονται πια τόσα πολλά παρασιτοκτόνα. Βλέπουμε όμως ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την άμυψη σπορά, διότι δεν μπορείτε να καταδικάσετε τον Μένο Βασίλειο για να ικανοποιήσετε τους δανούς και τον υδροφόρο ορίζοντά τους. Τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητές από διάφορες πολιτικές ομάδες. Η κυρία Τίσεν για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι συνάδελφοί μας εργάστηκαν σκληρά για μια συμφωνία η οποία αξίζει να υποστηριχθεί διότι και φιλόδοξους στόχους έχει αλλά και διότι η γεωργία μπορεί να παραμείνει σε συμφωνία με την οικονομία και να διατηρηθεί και η ανταγωνιστικότητά της. Συμβασμός σημαίνει ένα δούνε και λαβίν. Με ορισμένα κριτήρια δεν είμαι απόλυτα σύμφωνη. Θα προτιμούσα ε, να ξεκινήσουμε με μια επιλογή και όχι με ε, μια επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου. Αλλά φαίνεται πως αυτό ήταν ε, ο μόνος τρόπος. Υπάρχουν θετικά σημεία. Οι χώρε μέλη διατηρούν ένα περιθώριο ελιγμών για, την, για τον καθορισμό της, των μειώσεων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίζεται σε τρεις ζώνες σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση. Η γραφειοκρατία μειώνεται και υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φυτοφαρμάκων. Οι χώρες μέλη λαμβάνουν την υποχρέωση να είναι πιο ε, ευέλικτες, επίσης να δημιουργήσουν ζώνες προστασίας γύρω από τα διάφορα ε, εσωτερικά ύδατα και να χρησιμοποιούν ε, με λελογισμένο τρόπο τα φυτοφάρμακα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές χώρες με μικρή επικράτεια. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτές τις μικρές χώρες και ελπίζω ότι ε, θα ενισχυθούν και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή τα φυτοφάρμακα. Εάν υπάρξει λογικός, δελογισμένος έλεγχος και εάν χρησιμοποιηθούν με επαγγελματικό τρόπο και λάβουμε και υπόψη ότι η γεωργία θα πρέπει βεβαίως να είναι ανταγωνιστική και διεθνώς. Εάν μπορούμε λοιπόν να κλώσουμε τους στόχους αυτούς, τότε θα έχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δρόμο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πως τα φυτοφάρμακα είναι αυτά, τα, τα, οποία έχουν επιτρέψει να αυξηθεί η ε, γεωργική παραγωγή έχουν ωστόσο επιπτώσει πολύ αρνητικέ για την υγεία και για το περιβάλλον. Γι' αυτό πέρα από την νομοθεσία που θα θεσπιστεί είναι επίση επίγον να δημιουργηθούν ε, μητρό επιδημιολογικά που να επιτρέπουν ε, να μετρά το αντίκτυπο των διαφόρων ε, ζυζανιοκτώνων ανάλογα με την εργασία των επαγγελματιών του κλάδου και των οικογενειών τους, χωρίς να ξεχνάμε και τους καταναλωτές των διαφόρων περιοχών. Σε ορισμένε περιοχές βλέπουμε την ε, ιδιαίτερα ταχεία αύξηση ορισμένων ειδών καρκίνου. Τα παιδιά των καλλιεργητών ε, και οι ίδιοι καλλιεργητέ ε, πλήττονται. Ε, πέρα από την υγεία θα πρέπει να μετρήσουμε τι επιπτώσει στο περιβάλλον. Γνωρίζουμε ήδη τι αρνητικέ επιπτώσει των χημικών προϊόντων στου υδροφόρου ορίζοντε και στα ποτάμια. Και γι' αυτό και θα πρέπει να μιλήσουμε για τι ζώνε σύνορα, αλλά δεν νομίζω πως είναι επαρκής αυτή η απάντηση. Η Κομισιόν σε αυτό το θέμα θα πρέπει να επαγρυπνεί ιδιαίτερος. Επίσης σήμερα παρατηρούμε μια αύξηση της διάβρωσης των γεών που μπορεί να αφισβητήσει την ε, γεωργική χρήση πολλών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επόμενες δεκαετίες. Η γονιμότητα αυτών των γεών μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά και είναι καλό. Αλλά θα πρέπει επίση να συνοδεύσει του ε, γεωργού σε μια απόπειρα μείωση και ίσω και κατάργηση των ε, ζυζανιοκτώνων. Ε, θα πρέπει να θεσπίσουμε καλύτερα του στόχου για να λάβουμε υπόψη τη σύνδεση ανάμεσα στην ποιοτική παραγωγή και, τους γεωργού, και τη γεωργία η αγρονομική έρευνα, η έρευνα στην αγροτοξικολογία, καθώς και η χρήση νέων μεθόδων παραγωγής θα πρέπει να σχετίζεται και με την παραγωγικότητα της κάθε περιοχής. Να σας θυμίσω ότι θα πρέπει να δούμε και το έργο Αύριο τα παιδιά μας θα μας κατηγορήσουν. Είναι μια ταινία που βγήκε πρόσφατα και θα πρέπει όλοι να τη δούμε. Αφορά αυτά τα θέματα. Αντρουσκά για 1,5 ε, λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ευρωβουλευτές που θεωρούν ότι η Συμφωνία Δεύτερης Ανάγνωσης είναι μια σωστή εξισορροπημένη λύση δεδομένης της περιπλοκότητας του θέματος. Ε, μας υποδεικνύει το δρόμο για περαιτέρω βελτιώσεις στον τομέα προς πιο αποτελεσματική και πιο για πιο αποτελεσματικά και ασφαλή προϊόντα για φυτοπροστασίες καθώς και είναι επαρκώς ευέλικτη ώστε να μην μας οδηγήσει στην απαγόρευση της χρήσης ορισμένων ε, ζυζανιοκτώνων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω την βελτίωση του αρχικού της αρχικής πρότασης της Κομισιόν που στόχο έχει την αποφυγή της επικάλυψης δοκιμών και μελετών και να προωθήσει τις δοκιμές ε, άνευ ε, πειραματόζων. Επίσης, ε, για τα στοιχεία για την προστασία των φυτών προχωρούν τώρα στη δική τους διαδικασία αναθεώρησης. Ακόμα και αν τα ζενιοκτώνα σε με χημικά ε, έχουν στόχο να είναι τοξικά και άρα η αξιολόγηση ασφάλειας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, θα πρέπει να γίνονται περιττές δοκιμές σε ζώα ή ότι η επιστημονική γνώση δεν μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπους που θα εντοπίσουν περαιτέρω περιτά στοιχεία και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των δοκιμών σε ζώα στο μέλλον. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη και η καταγραφή των νέων γεωργικών ζυζανιοκτώνων ή προϊόντων φυτοπροστασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει χιλιάδες ζώα σε πολύ συχνά επικαλυπτόμενες δοκιμές. Ο κύριος Ρούτοβιτς έχει το λόγο. pani przewodnicząca! drodzy państwo! pestycydy są środkami groźnymi dla zwierząt i środowiska. chciałbym <laughs> προϊόντα πολύ συχνά είναι επιβλαβή για τα ζώα και για το σε πολλές χώρες όλα τα αποθηκεύονται σε πολύ για το περιβάλλον και για τους ανθρώπους. χωρίς τη βοήθεια της δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα η εξισορροπημένη χρήση των ζυζανιοκτώνων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε τους χρήστες καθώς και να τους βοηθούμε στις ε, διάφορες, μέσω διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών. Τα ζυζανιοκτώνα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται σε ε, υπερβολικές ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες και κυρίως αυτό αφορά τους μικρούς χρήστες οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη ε, αγροτεχνική γνώση για τα ζυζανιοκτώνα. Είναι πολύ σημαντικό το πώς τίθεται σε εμπορία τα ζυζανιοκτώνα. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επιστημονικές έρευνες από αυτόν και να εστιάσουμε στις δραστηριότητες που καθιστούν την χρήση συζανιοκτώνων πιο περιορισμένη και ω εκ τούτου και πιο περιορισμένη την επιρροή του στην υγεία και στο περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέγκερ για αυτή την έκθεση και να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό πω η οδηγία αυτή θα έχει νόημα αν αυτέ οι οδηγίε θα έχουν νόημα αν πραγματικά εφαρμοστούν στην γεωργική πρακτική. Είμαστε υπέρ αυτή τη οδηγία. Λεπτά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία για την υπεύθυνη χρήση ε, φυτοφαρμάκων ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και οι δύο οδηγίε που συζητάμε εδώ είναι σημαντικέ. Ε, η προστασία τη υγεία είναι ένα ε, βασικό δικαίωμα των ανθρώπων. Εμεί θέλαμε μια πιο ισχυρή ε, απόφαση στο τέλο, ένα πιο ισχυρό αποτέλεσμα. Παρ' αυτά θα συμφωνήσουμε. Για την άλλη μεριά θα πρέπει να μην ξεχνάμε τι αντιδράσει του αγροτικού τομέα και τη βιομηχανία παραγωγή των φυτοφαρμάκων αυτών. Εμείς θέλουμε να προσπίσουμε καλύτερη προστασία και των φυτών και των ζώων και να υπάρχουν καλύτερα προϊόντα. Ο κρατικός τομέας μας επέκρινε και είπε ότι θα εξαφανιστεί το ίμιση του τομέα αυτού. Αυτό δεν είναι βέβαια αληθές. Πάνω από 90% των προϊόντων θα εξαφανιστούν, είπανε. Δεν είναι ζωστό αυτό. Δεν είναι αληθές. <clears throat> Γιατί το λεγόμενο phasing out θα διαρκέσει πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια απαγόρευση πόρων οι οποίοι έχουν επιβράσει στο ορμονικό μηχανισμό που είναι καρκινογόνο κλπ. Με όλο το σεβασμό στην αγροτική βιομηχανία θα ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ίσως και ένα έκτακτο σχέδιο για να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο αγροτικό τομέα. Χρειαζόμαστε ειλικρινό συμβασμό μεταξύ της οικολογίας και της γεωργίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό η συνάδελφος Μαριλού Μακτόναλτ έχει το λόγο. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα περιβαλλοντικής πολιτικής που βελτιώνει και τη ζωή των πολιτών. Αλλά έχουμε και παραδείγματα προς αποφυγή, κατά τα οποία έχουμε γραφειοκρατικά παραδείγματα τα οποία μπλοκάρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών και δυστυχώς θεωρώ ότι αυτό το νομοθέτημα εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία. Θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν εννοώ την βιομηχανία, εννοώ τους γεωργούς. Όπως τα είπε και η προλαλήσασα, οι γεωργοί προβληματίζονται και ε, ενδιαφέρονται όπως οποιοδήποτε για την ανθρώπινη υγεία. Δεν υπάρχει η εθνική τεκμηρίωση τόσο ώστε να βοηθεί και η ε, οικονομία μας. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη επομένως όλα όσα θα βοηθήσουν την ε, οικονομία μας εάν γίνει εφαρμογή αυτήν της δέσμης μέτρων η οποία έτσι όπως είναι τώρα θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα καλόπιστη είναι η θέσπιση αυτής της νομοθεσίας όμως αυτή τελικά πρόκειται την Ήπεθρο να την βλάψει με μια αυστηρή νομοθεσία η οποία θα πλήξει την ήδη πλησόμενη τάξη των γεωργών. Και ξέρετε στην Ιρλανδία όλοι οι γεωργοί ομόφωνα απορρίπτουν αυτές τις προτάσεις. Προσοχή, λάβετε υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πολιτών, των γεωργών τα οποία δεν ωφελούνται. Έχουμε μία θέση από τον τριγωνικό διάλογο που βελτιώνει την αρχική πρόταση, αλλά ε, ό,τι και να κάνουμε δεν καλύπτουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Νίλς Λόντκρεν, παρακαλώ. Ja, fru talman, det är ovant för en övertygad EU-skeptiker som jag att... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε αυτός ο σκεπτικισμός που υπάρχει σχετικά με την έκθεση δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε. Αυτό θα σήμαινε ότι οριοθετούμε για το πρόβλημα του περιβάλλοντος και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της αγοράς μας επίσης προσπαθούμε να δράσουμε κατά τέτοιο τρόπο ούτω ώστε να βρούμε μη γραφειοκρατικές λύσεις. Οι πρόταση που έχουμε μπροστά μας θέλουν να μειώσουν την ε, γραφειοκρατία και να οδηγήσουν σε αυστηρούς ελέγχους ε, ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται επικίνδυνα θα πρέπει να ελέγχονται λέγεται. Ε, αυτή είναι η πρόταση. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ σωστό. Επίσης ε, τα διάφορα κράτη μπορούν, άμα ε, θέλουν, να απαγορεύσουν από μόνα τους κάποια προϊόντα. Από την άλλη μεριά, ορισμένα φυτοφάρμακα μπορούν να ε, χρησιμοποιούνται, να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι που είπαν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος εάν εισαγάγουμε πιο αυστηρούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τότε ίσως θα αγοράζονται αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Απ' την άλλη μεριά δεν μου φαίνεται ότι αυτό το επιχείρημα είναι πολύ βάσιμο για να καταψηφίσουμε. Πρέπει να υπερψηφίσουμε την συμβαστική πρόταση. Reagan, Πρόεδρος, δεν βλέπω τον συνάδελφο Τόμας Βάις. Η Φωνσάς Γκοστέτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να συγχαρώ το, την εισηγήτρια και να χαιρετήσω τη συμφωνία που εξευρέθη χάρη στην εξαιρετική εργασία της εισηγήτριας αλλά και της υποβοήθησης από την Κομισιόν και το Συμβούλιο γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία που είναι ισορροπημένη και που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων δηλαδή η προστασία της υγείας του καταναλωτή αυτού του καταναλωτή που ανησυχεί από τη στιγμή που αρχίζουμε και μιλάμε για ζενεοκτώνα, που ανησυχεί όταν ακούει για κατάλοιπα των ζενεοκτώνων που μολύνουν τα φρούτα, τα δημητριακά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν κατάργηση των καρκινογόνων και τοξικών ουσιών, πολύ σημαντικό, προστασία της περιβάλλοντος και της ε, ε, βιοπικιλότητας, προστασία των μελισσών, των γεών, των υδάτων και, αλλά και των γεωργών που είναι και οι ίδιοι ε, ε, άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη χρήση αυτών των ζενιοκτώνων και με ικανοποίηση θα δουν την εναρμόνιση της ε, νομοθεσίας, την απλοποίηση της διαδικασίας, τη δυνατότητα πάντοτε να μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένε ουσίες που χρειάζεται για να ε, μπορεί να κάνει γεωργία, αλλά την οποία γεωργία θέλουμε πια σήμερα να είναι βιώσιμη. Και έπειτα υποχρέωση της χημικής βιομηχανίας να εξελιχθεί, να βρει εναλλακτικέ λύσεις. Αυτή τη χημική βιομηχανία την οποία χρειάζεται η γεωργία, αλλά που πρέπει οπωσδήποτε να βρει εναλλακτικέ λύσεις. Με το κείμενο αυτό δεν θα μπορούμε πλέον να συγχαίουμε τις έννοιες του κινδύνου και του ρίσκου. Τα ζυζενιοκτώνα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν ε, τρόποι για να ορίσουμε αν αυτοί, αυτά αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για τον καταναλωτή, την υγεία και το περιβάλλον. Καλή κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου, κατάρτιση του ευρέως κοινού, αλλά και θα τελειώσω λέγοντα ότι πρέπει οπωσδήποτε να εναρμονιστούν οι έλεγχοι των εισαγωγών. Γιατί δεν μπορούμε να πετούμε πράγματα από του γεωργού μα, αλλά να ξεκολουθούμε να εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα που δεν σέβονται τη δική μα νομοθεσία. Γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνο αθέμητου ανταγωνισμού. Σα ευχαριστώ. λεπτό, Madam Chairman, thank you. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγχωρήστε με που είμαι τσαγανιασμένος, αλλά η Air France που δεν μου βρήκε στην πτήση μου θέση και βρήκε στην επόμενη. Θυμάμαι τον Βλαντιμίρ Ήλιτς Λένιν που είχε πει ότι το χειρότερο είναι καλύτερο. Γιατί σε όλη μου αυτή την θητεία βλέπω τα πράγματα πηγαίνουν στο χειρότερο. Όμως το χειρότερο είναι καλύτερο και ε, κατ' εμέ είναι καλύτερο διότι ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει πόσο κακή είναι η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το φαγητό που τρώνε, για το εισόδημά τους, για τη ζωή τους. Γιατί αυτό θέλει να προβάλλει το κόμμα μου. Τίποτα δεν κάνει για τους κινδύνους, ούτε για τις βλαβερέ συνέπειες των ε, φαρμάκων αυτών ε, και επομένω δεν αποδίδει αυτή η νομοθεσία, πέθει στο κενό, τελικά θα πλήξει την παραγωγή, θα σπρώξει στο να φαλυρίσουν οι γεωργοί και όλα θα γίνουν χειρότερα. Επομένως, εμείς καταψηφίζουμε. Ε, ε, πάντως, ε, ε, όταν ε, προχωρήσετε ένα τέτοιο νομοθέτημα, ελπίζω να φύγει η χώρα μου την Ένωση. Δύο λεπτά τώρα η κυρία Κόρμπη. Dank Και εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές αλλά και τους χιώδες συγητές και πιστεύω ότι αυτός ο συμβασμός είναι ένα θετικό βήμα ούτως ώστε να γίνει κάτι για τη γεωργία, κάτι που το χρειάζονται όλοι πάρα πολύ διότι όλα αυτά τα φάρμακα είναι πολύ σημαντικά ούτως ώστε να προλαβαίνουμε ε, τις ασθένειε που πλήσουν την ε, παραγωγή. Επίση, θα πρέπει να φροντίσουμε και το περιβάλλον, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την υγεία την ανθρώπινη. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο ε, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ της συμβατική γεωργία και της βιολογική γεωργία. Έχουμε τώρα τρία μέτρα εδώ σημαντικά τα οποία προβλέπονται. Πρώτα-πρώτα τι γίνεται για τα ιδιαίτερα πήγαινα χημικά, θα απαγορευτούν και προβλέπονται όμως κάποιες παρεκκλήσεις εάν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εναλλακτικέ. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα θα δημιουργήσουμε στη Γεωργία. Επίσης προβλέπονται κάποια κίνητρα ούτως ώστε να γίνει χρήση των σωστών φαρμάκων από τους ε, μικροπαραγωγούς, από τους κυπουρούς ε, και για τα απορροκυπευτικά όπως οι Οι πόλεμοι πάντως φοβούνται ότι θα απειληθεί αυτή η μικρή κλίμακα καλλιέργεια. Όμως δεν είναι έτσι, διότι προβλέπονται ε, ειδικοί πόροι οι οποίοι πρόκειται να ενισχύσουν την έρευνα για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Επίσης προβλέπεται το πώς θα μειωθούν ε, οι, με κάποια έρευνα πώς θα μειωθούν οι κίνδυνοι για επικίνδυνα προϊόντα ε, και πώς δεν θα παραβλαβεί το περιβάλλον ευαισθήτων περιχών όπως ας πούμε ε, κάποιες γειτονές βρίσκεται ένα σχολείο. Οπότε τώρα θα κάνουμε καλό και στην υγεία και στο περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα όλα τα χημικά αυτά να, τα επικίνδυνα να απαγορευτούν γιατί νομίζω ότι είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χαίρεται σήμερα για τα όσα πέτυχαν η Κομισιόν, το Συμβούλιο και φυσικά η σε αυτό το θέμα των ε, φυτοφαρμάκων. Φυσικά μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερη πίεση, πολύ ευαίσθητο το θέμα, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Πρόκειται για ένα νομοθετικό, ε, μια νομοθετική δέσμη που συνδυάζει και, και περιβάλλον και καινοτομία με και έρευνα αντί να τα αντιπαραθέτει όπως συχνά συμβαίνει. Πρόκειται για πολλά χημικά προϊόντα τα οποία αναμφίβολα παίζουν ε, σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση των ζωνίων, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που καταγγέλουν αποφευκταίους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και κυρίως να πούμε για τους γεωργούς που αυτοί περισσότερο ε, εκτίθενται στους ενδοκρινικούς διαταράκτες και στα και, έχουμε περίπου 1.200.000 ε, θανάτους ε, ετησίως ε, σε τάξη των γεωργών λόγω αυτών των ζυζανιοκτώνων να δούμε τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ε, ελπίζουμε πως έτσι θα μιλήσουμε για μια φιλόδοξη πολιτική, ρεαλιστική και πραγματικά πολύ σύγχρονοι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν και περιμένουν από εμά να σταματήσουμε τη χρήση αυτών των επικίνδυνων ζενοκτώνων. Ρεαλιστική διότι γίνονται σεβαστοί οικονομικοί κύκλοι ζωή τα δύο τρίτα μπορούν να τεθούν στην αγορά και υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση κάθε 10 χρόνια. Άρα λοιπόν η βιομηχανία θα πρέπει να ανησυχεί και είναι σύγχρονο αυτό, αυτή η δέσμη γιατί το θέμα των Ζανιοκτώνων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο με την Ευρώπη, για την Ευρώπη λιγότερα αλλά καλύτερα παρασιτοκτόνα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Κούτσνιουκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, όταν ε, μιλάμε για την ε, εφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και των ε, φαρμάκων προστασίας των φυτών, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, δύο στάδια στην χρήση χημικών ουσιών. Καταρχήν, δηλαδή, η εισαγωγή για την εμπορία τους και την εφαρμογή του. Δεν συζητάμε όμω το θέμα τη απόσυσης των προϊόντων αυτών και τη ανακύκλωσή του. Στην Πολωνία βλέπουμε να υπάρχει ανάγκη να υπάρχει έντονη ανάγκη οικονομική ενίσχυση για το τρίτο αυτό στάδιο, για να μπορούσαν δηλαδή οι τοπικές αρχές να αποσύρουν και να ανακυκλώσουν ή να καταστρέψουν αυτές τις ουσίες. Επίση θα ήταν χρήσιμο να διαβεβαιώσουμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των προϊόντων αυτών στι αγορέ τους. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω την ε, πεποίθησή μου ότι οι λύσεις που συζητάμε σήμερα οδηγούν σε επίπεδο δύο παιχνίς για όλους τους ε, γεωργούς. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Η κυρία Ντεγκόμεζο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προτάσει τη έκθεση αυτή κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση και συγχαίρω του συγγετρίε. Εάν, όπω είπε η Κομισιόν, τα φυτοφάρμακα αφορούν κυρίω την κοινή αγροτική πολιτική, παρ' αυτά μια τέτοια οδηγία θα πρέπει να έχει σαν στόχο μια νομική βάση που θα εστιάζεται στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Αλλιώ έχουμε απλώ ένα θέμα αναρμόνιση αγορά ή αναγνωστικότητας. Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα από την Γουαδελούπη και την Μαρτινίκα, όπω στη Μαρτινίκα το 20% των εδαφών το 20% δηλαδή όλη τη επιφάνεια τη νήσου, ενό εκατομμυρίου και κοινωνικών κινημένων έχουν καταστραφεί από ουσίε που δεν είναι γνωστέ. Και αυτό αφορά όχι μόνο τα εδάφη, αλλά επίση και τα υπόγεια ύδατα και τις, ε, ε, τους ακρογιαλιές. Εις βάρος της οικονομίας μας εάν δεν ακόμα πολύ αργά, να γνωρίσει παρακαλώ το Κοινοβούλιο την περίπτωση της Μαρτινίκας που την ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Γάλλοι που λέγεται θα πρέπει να απογραφθούν αμέσω η χρήση των χημικών ε, λιπασμάτων και θα πρέπει γι' αυτό να χρησιμοποιούμε μόνο ε, βιολογικά στοιχεία. Παρακαλώ, Άλλη Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα των μελιστών. Θα πρέπει επίσης να ε, παγρυφνεί το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα ε, προϊόντα ελεύθερης συναλλαγές που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε για τη χρήση εκεί των ε, φυσοφαρμάκων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ένα λεπτό και ζησινότητα. What we in here is a desire to protect health, but we should remember that... Εκτός από την υγεία, να θυμηθούμε ότι η υγεία μας βασίζεται στο, στην τροφή που παράγουν οι γεωργοί και εγώ προέρχομαι μια τέτοια οικογένεια γιατί έχουμε ε, τα διάφορα έντομα αλλά και διάφορα παράσιτα τα οποία πλήσουν την παραγωγή κάτι το οποίο στην Ιρλανδία έχει πλήξει ιδιαίτερως ε, την παραγωγή και όμως αυτό ήδη ε, γίνεται το εξής έχουμε δημοσιεύσεις για παραγωγή μεταλλαγμένων πατατών, κάτι το οποίο ε, θεωρείται ως αντίδραση στα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας λένε επίσης ότι το DNA των φυτών πρόκειται να διατραχθεί και επομένως τώρα περισσότερο ποτέ θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Φερδινόντε Ροσινέλ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, μετά από τον τρεμερή διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν, το κείμενο που υιοθετήθηκε στι 18 Δεκεμβρίου για το δέσμη για τα παρασυντοκτόνα φαίνεται να είναι ισορροπημένο. Λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των γεωργών και την απαραίτητη προστασία του περιβάλλοντο καθώ και των προστατευόμενων ζωνών. Χαίρομαι λοιπόν, χαίρομαι για το αποτέλεσμα που θα επιτρέψει στου γεωργού να συνεχίσουν την οικονομική του δραστηριότητα δραστηριότητα χωρίς να τιμωρηθούν από την απόλυτη κατάργηση των παραστοκτώνων και των, φυτο... και των προϊόντων φυτοπροστασίας που αυστηρά θα πλαισιωθούν. Να θυμίσω ότι η παραγωγή ε, ε, των ε, λαχανικών και των εσπεριδοειδών στην Νορμανδία, στην την περιοχή που αντιπροσωπεύω. Εδώ και καιρό ακολουθούν αυτού του κανόνε και χαίρονται που ολοκληρώνεται έτσι μια περίοδο μεγάλη επιβεβαιότητα λόγω τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ και των απειλών που βαραίνουν τον προπολογισμό. Εμεί είμαστε υπέρ των εργαλείων εργασία των γεωργών και το αναλύω του ρόλου του στην κοινωνία που είναι να θρέψουν τον πληθυσμό αλλά και να προστατεύσουν το, τις της ΓΕΕΣ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η κοινή λογική να κερδίσει εδώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ανεβάσει βέβαια. κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αύριο θα ψηφίσουμε για νέους διαγωνισμούς στο θέμα των φυτοφαρμάκων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, κινεί πάρα πολύ τους πληθυσμούς. Αυτό αντικατοπτρίζεται και συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Όλοι θέλουμε να έχουμε υγιή και φρέσκα τρόφιμα από τις περιφέρειές μας σε τιμές αποδεκτές χωρίς κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Το αποτέλεσμα που επιτεύχθη στον τριμερή διάλογο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Ο νέος κανονισμός για τα φυτοφάρμακα αποτελεί σημαντική πρόοδο για περισσότερη προστασία του ε, κατανοητή και της υγείας. Καθορίζοντας όμως τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν ε, επιστημονικά κριτήρια και όχι πολιτικά δογματικά κριτήρια σε σχέση με το πρώτο αποτέλεσμα ε, είναι μεγάλη πρόοδος το αποτέλεσμα του τριλόγου γιατί αφορά όχι πια το 80% των προϊόντων αλλά εκείνους τα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Και έτσι θα έχουμε αρκετά φυτοφάρμακα στη ε, διάθεσή μας για να μπορούμε να καλλιεργούμε τα ε, διάφορα προϊόντα σωστά στην έγκριση των ε, φυτοφαρμάκων δεν θα έχουμε στο μέλλον 27 διαφορετικές υπηρεσίες εθνικές, αλλά τρεις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Εκεί θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τις εγκρίσεις τους. Ο νέος κανονισμός για τα φυτοφάρμακα μας οδηγεί στην απαραίτητη εναρμόνιση και στον τομέα αυτών. Έτσι έχουμε ένα ομοιόμορφα υψηλό επίπεδο ε, προστασίας χωρίς να διακυβεύουμε την αηφόρο καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έχουμε πραγματική ιστορική αγορά, ενιαίο όρους ανταγωνισμού και μεγάλη πρόοδο για την προστασία της υγείας. Σημαντική πρόοδος και για τους κατανοητέ και για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά. Τατιάνα Σαρμπού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν με τρόπο αποτελεσματικό με αυτές τις κατάλληλες δόκιμες πρακτικές τόσο ώστε να γίνεται παραγωγή τροφίμων με παράλληλη προστασία του καταναλωτή αλλά και του περιβάλλοντος. Η δε μείωση και περιορισμός των κινδύνων από αυτά τα φυτοφάρμακα πρόκειται να βοηθήσει ούτως ώστε να έχουμε μια βιώσιμη γεωργία μεγάλη χρήση τέτοιων, εκτεταμένη χρήση τέτοιων ε, φαρμάκων ε, γίνεται ε, λόγω της εξάρτησής μας από αυτά τα χημικά προϊόντα τα οποία μέχρι ενός σημείο χρειάζονται για μια αποτελεσματική παραγωγή όμως μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη δημοσία υγεία πολλά κρατημέλη αλλά και η Ρωμανία έχουν πρόβλημα όσον αφορά κάποιες ασθένειες που χτυπούν την παραγωγή και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα, αυτά τα χημικά. Χρειάζεται όμως μια σωστή διαχείριση ε, του κινδύνου και έτσι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτά τα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη την προστασία και του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις αρτησίες μας από αυτά τα χημικά. Όλα αυτά τα ζυζάνια, όλα αυτά τα οποία πλήσουν την παραγωγή στην Ρωμανία είναι τόσο πολλά τα οποία μας αναγκάζουν να προσφύγουμε σε τέτοιες λύσεις. <coughs> Έχουμε και ψεκασμούς οποίος εκτεταμένος, όμως όταν ισχύσει αυτή η νομοθεσία θα γίνεται υπό όρους ο ψεκασμός και έτσι θα προστατευτεί το περιβάλλον. Χαίρομαι που προέκυψε αυτός ο συμβιβασμός, ένα συμβιβασμός που βρήκε σύμφωνα στις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετή ποσότητα τέτοιων χημικών, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά και θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτά. Όλγα Κράμα. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Τα φυτοφάρμακα ήταν και εξακολουθούν να είναι σημαντικά μέσα χρήσης από τους γεωργούς. Χρειάζεται η γεωργία να προστατεύσει τις καρδιές μας ε, επιφάνειες και να εξασφαλίσει την ε, τροφοδοσία του πληθυσμού. Πολλές φορές ε, το θέμα αυτό συζητιέται πολύ συναισθηματικά, θα πρέπει όμω να σκεφτούμε και να δράσουμε ορθολογικά. Οι επιπτώσει τη αρχική θέση του Κοινοβουλίου θα ήταν μοιρέ. Η γενική απογόρευση δηλαδή των φαρμάκων θα οδηγούσαν σε λιγότερη απόδοση και άρα σε αυξημένες ε, τιμές ε, τροφίμων. Χαίρομαι λοιπόν που στην τριμερή διάλογο πετύχαμε μία λύση η οποία μπορεί να είναι αποδεκτή. Είναι καλό που διατηρήσαμε τις τρεις αυτές ζώνες αλλά με σημαντικές εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη. Η τολμηρή λύση ήταν βέβαια διαφορετική. Εκτός από τις αποδεκτές ε, συμβαστικές λύσεις θα πρέπει να έχουμε μία οριστική να μην προτρέξουμε μάλλον μια οριστική ε, δυνατότητα ορισμού των ενδοκρίνων ε, ουσιών. Θα πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα, αλλιώς ε, θα καταπατήσουμε την αρχή της πρόληψης και επίσης λυπούμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμφωνίας που επιτεύχθη τώρα. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Γιάννος Ποτσεκόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα βάζω τελευταίες πινελιές σε αυτό το νομοθέτημα ούτω ώστε ε, να διευθετηθεί το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Είναι εύστοχος και δίκαιος ο συμβασμός ούτω ώστε θα υπάρξουν τώρα κάποιοι περιορισμοί και έτσι θα προστατευτεί η δημόσια υγεία χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξει κάποιος φραγμός στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Βεβαίως και θα πρέπει να προσέξουμε ποιο είναι το κόστος αυτών των μέτρων γιατί θα πρέπει να παραμείνει στην διεθνή σκηνή ανταγωνιστική γεωργία μας. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο ήδη προελέχθη. Θα πρέπει να είναι ψηλά ο πύχης όσον αφορά τους ε, γεωργούς, όσον αφορά τους εργαζόμενους στη γεωργία. Όμως θα πρέπει οι ίδιοι αυστηροί κανόνες να ισχύσουν και για τις εισαγωγές. Για να μην γίνουμε αντιπαραγωγικοί με το νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Τζιμάλιστερ. President, I do not accept that Πρόεδρε, δεν δέχομαι ότι έχουμε ε, ισορροπημένη δέσμη για αυτό το θέμα. Εδώ τονίζονται δύο παράλογα πράγματα. Καταρχήν, η παράλογος τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί καμιά αξιολόγηση προχωρά στην απαγόρευση διαφόρων ε, παρασιτοκτόνων χωρί να ενδιαφέρεται για το ότι δεν υπάρχουν ε, υποκατάστατα και ότι η εγχώρια παραγωγή τροφίμων θα υποφέρει ιδιαίτερα στα δημητριακά και στα λαχανικά και επιβάλλουμε έτσι ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές από χώρες που καρφάκι τους καίγεται για όλα αυτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, εδώ γίνεται πολλής λόγος για επιστήμη. Μα τι είδους επιστήμη είναι αυτή που δεν υποβάλλει τον εαυτό της σε πραγματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων. Η δεύτερη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι αυτός της χώρας μου ιδιαίτερα που επηρεάζεται ίσως περισσότερο από αυτές τις προτάσεις και που έχει ε, μπει, είχε δεχτεί την ειδική πλειοψηφία ε, στο Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Εδώ που φτάσαμε μάλλον δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε και λόγω στη, της ανοησίας του να δεχτούμε την, την, την ειδική πλειοψηφία βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και ωστόσο ορισμένοι λένε για τη Λισαβόνα και λένε ότι όλα είναι και περισσότερο θα πρέπει να γίνονται, λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αυτές οι αποφάσεις, η ειδική πλειοψηφία. Δύο λεπτά, ο κύριος Ζήπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται νομίζω για μια ισορροπημένη συμβαστική λύση και θα την υποστηρίξω και θα ήθελα από τη ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν. Όπως ακούσαμε και στη συζήτηση, ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση που έγινε προηγουμένως, αλλά μπορέσαμε να επιτύχουμε να ε, προστατεύσουμε όπως θέλαμε βάσει του κανονισμού. Η Ευρώπη έχει έτσι μία από τι πιο προηγμένε θεσίες για τα φυτοφάρμακα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν σημαντικό να επιτευχθεί μία ισορροπία μεταξύ τη προστασία, τη υγεία, τη εσωτερική Αγορά και του περιβάλλοντο, αλλά και να υπάρχει και μία ισορροπία μεταξύ αυτών των στόχων. Και επιτεύχθηκε εκεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν να λάβουμε υπόψη αυτέ τι διάφορε αρχέ ότι παραδείγματο χάρη ότι όλα θα πρέπει να βασίζονται πάνω σε επιστημονικά στοιχεία και όχι σε συναισθήματα. Και δεύτερον, βασιζόμαστε στο κίνδυνο, στο ρίσκο και όχι στον άμεσο κίνδυνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω για την εφαρμογή των ε, μέσων αυτών, των αποφάσεων αυτών. Επίσης θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι κατά την εφαρμογή δεν θα ωφεληθούν ε, τις αγωγές εις βάρος της εδοκοινωτικής παραγωγής. Πολλά πρέπει να κάνει η Κομισιό εδώ, αλλά νομίζω μια που λάβουμε υπόψη μας ισορροπημένα αυτές τις αρχές θα μπορέσουμε να δεχτούμε και να συμβαστούμε με το συμβιβασμό. <clears throat> Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα της προστασίας των υδάτων. Εκεί θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για την ε, επικουρικότητα γιατί δεν μπορούν όλα να ε, συγκρίνονται μεταξύ τους η Γερμανία με τη Μάδια, με την Ελλάδα ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται επίσης με τα φυτοφάρμακα μέσα στα πλαίσια του Natura 2000 και εκεί τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα της σωστής εφαρμογής γενικά δηλαδή ένα συμβασμό που μπορούν νομίζω να επομισθούν όλοι Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Πόπταν ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και πρώτα πρώτα να συγχαρώ τους συνεισηγητές. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας πολύ, οπότε και θα σταθώ στην έκθεση της κυρίας Κλάς. Έχουμε μια οδηγία που θεσπίζει αυτό το σύστημα των πιστοποιητικών τα οποία θα πρέπει να χορηγούνται σε κάποιους καλλιεργητές και βέβαια βασίζονται αυτά τα πιστοποιητικά σε σύστημα αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης με αυτή την οδηγία συνεχίζουν ενισχύει οι εθνικές διατάξεις. Βέβαια θα πρέπει να ανθεωρηθεί ε, αυτή η πρόβλεψη και να υπάρξει ρύθμιση σε ευρωπαϊκό, ενωσιακό επίπεδο. Θα πρέπει πάντως και οι δοκιμές να την χάνουν αναγνώρισης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ιδίως όσον αφορά τις ε, παραμεθόριες περιοχές και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει όσον αφορά ε, τη, τη δασική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ως Ευρωβουλευτής Παρακολούθησα φυσικά αυτή την νομοθεσία με πολύ ενδιαφέρον και πολύ ανησυχία. Μιλάμε για πολύ ιδιαίτερο θέμα και για τη δική μου χώρα, τις κάτω χώρες, την Ολλανδία, όπου πραγματικά επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τα ζενοκτώνα. Αντίθετα από αλλού στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να χρησιμοποιήσουμε προζώνες προστασίας ε, μαζί με τα δίπλα μάλλον στα κανάλια. Μια τέτοια προσέγγιση θα καθιστούσε τις ε, κανονικές μεθόδους παραγωγής αδύνατες. Ε, εμείς εξάλλου έχουμε ανέκαθεν προωθήσει τις μικρές παραγωγές, τους μικρούς λαχανόκηπους και γι' αυτό και είναι πολύ καλό για μας ότι αυτό αυτός ο συμβιβασμός είναι εξαιρετικά πιο λειτουργικός από ότι αυτός που είχε προτείνει η κυρία Μπράγκερ στην Επιτροπή και γι' αυτό και μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Έχουμε καλά μεταβατικά μέτρα που σημαίνει πως η βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει την κοινοτομία για να βρει <coughs> αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις. Και ε, φυσικά τονίζουμε την ανάγκη για την χρηματοδότηση των γεωργών ώστε να μπορέσουν να περάσουν από αυτή τη δύσκολη περίοδο και να... τα μέτρα αμοιβαίας αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ πιο πρακτικά. Δύο παρατηρήσεις ακόμη. Καταρχήν η, προσ... η εισαγωγή εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να βρούμε μια αποτελεσματική ισορροπία ανάμεσα στι υγιεί ανάγκε, στι ανάγκε μάλλον για την υγεία και τι ανάγκε για το περιβάλλον, αλλά θα γίνει με τι εισαγωγέ. Μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, τέτοιου είδου θέματα τα οποία ανήκουν στον ανταγωνισμό ε, μπίπτουν μάλλον ε, στον ανταγωνισμό μπορεί να θυγούν και μπορεί να σημαίνει αυτό προβλήματα για τις αγωγές. Πολύ σημαντικό το θέμα. Να ευχαριστήσω την, ε, την και την κυρία Ένικοτα Ταπισέπιες που συνέβαλε ιδιαίτερα αλλά είναι κάτι στο οποίο επιμένουν οι Γεωργοί αυτό. Κάτι για το οποίο θα πρέπει να βρει λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ασφάλεια των ε, τροφίμων είναι ένα σημαντικό στόχο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ε, ο συμβασμός που έχουμε δεν είναι καλός γιατί οι Ούγγροι βουλευτές δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τον συμβασμό αυτό γιατί θα ήταν σε βάρος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Ο διακανονισμό αυτός για τις ζώνες είναι τεχνητός και είναι κατά της αρχής επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο Ολλανδός ε, συνάδελφος προηγουμένως, δεν επιτευχάνεται εδώ η απαραίτητη ευελιξία και αυτό είναι εις βάρος της ε, Ευρωπαϊκής Γεωργίας γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος, αυξάνεται ε, ο κίνδυνος της δυνατότητας αντίστασης των διαφόρων οργανισμών και όπως ελέγχθη δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εισαγωγές και γι' αυτό, αυτό ε, οι οδηγίες οδηγούν σε τεράστιο κίνδυνο και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ε, θα οδηγήσουν στο να μην χρησιμοποιούν αυτά και θα έχουμε γενικά τροποποιημένου οργανισμού που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Μαγκίνε, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι έδεξαν αυτές τις δύο σημαντικές εκθέσεις από όσα ακούσαμε απόψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχο στη θέση σε εμπορία αλλά και χρήση αυτών των χημικών. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν αυστηροί κανόνε για τα κατάλοιπα, για τα είδη διατροφή. Οπότε ούτε η μεν ούτε η δε από όσου επικρίνουν έχουν δίκιο. Ε, και επίση αυτοί που λένε ότι τώρα θα φέρουν μια τραγωδία, μια καταστροφή αυτά τα νομοθετήματα. Τώρα, ε, ανησυχούμε αυτό που είπε ο κύριος Δήμας. Είπε ότι ο κόσμος ανησυχεί για αυτά τα ζενιοκτώνα. Ναι, ανησυχεί. Το θέμα είναι πόσο δικαιολογημένα ανησυχούν και η Κομισιόν τι έκανε ούτως ώστε να εξηγήσει ε, στους παραγωγούς ότι προσπαθούμε να θεσπίσουμε κάποιους κανόνες για να έχουμε ε, υγιεινά τρόφιμα και ε, η καλή χρήση αυτών των χημικών γιατί το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την χρήση και θα χρειαστεί και από τα μέγιστα όρια κατάλοιπων. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι Γεωργοί. Έχουμε 22 ουσίες οι οποίε πρόκειται να απογραφτούν σε Ιρλανδία και σε Ηνωμένο Βασίλειο που ο κόσμος ανησυχεί για τις πατάτες και για τα σιτηρά. Το θέμα είναι η, τα, η, παραγωγή αγροχημικών θα ανταποκριθούν, θα μπορέσουν να παραγάγουν καλύτερα προϊόντα. Έχει απαντήσει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει εναλλακτικέ λύσει. Αυτά να σα απασχολήσουν γιατί εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε την παραγωγή μα όσον αφορά σιτηρά και πατάτε. Τώρα για τις εισαγωγές δώστε μου 5 και να σας εξηγήσω αυτό το σημαντικό θέμα γιατί εάν θέλει η Κομισιόν να βοηθήσει ε, τους παραγωγούς ειδών διατροφής μπορούμε κάτι να κάνουμε αλλά είναι απαράδεκτο η Κομισιόν να λέει απαγορεύουμε στην Ευρώπη αυτά τα χημικά αλλά μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτοί οι οποίοι μας ε, πουλάνε είδη διατροφής που εισάγουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να απαντήσετε πάνω σε αυτό απόψε. Σας ευχαριστώ. Δύο λεφτά για κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την εκθέση Μπράιερ. Ξέρουν οι Γεωργοί ότι τα αυτά τα φυτογενομικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο τόσο στη υγεία και περιβάλλον να μην παραβλάπτονται. Παρ' όλα αυτά αυτή τη στιγμή όλος ο κλάδος έχει προβληματιστεί γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταλαβαίνει Ποιε θα είναι οι συνέπειε από αυτά τα νομοθετήματα, Υπάρχουν κάποιε αξιολογήσει για τι επιπτώσει. Ήδη έχουμε ενδείξει για το ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσουμε τις ασθένειες που πλήσουν την παραγωγή κυρίως όσον αφορά ε, κάποια είδη που υπάρχουν στη Μεσόγειο όπως κάποια δικοσμητικά φυτά και άλλα κυπευτικά προϊόντα Έχουμε κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις βέβαια για να τον αυτό το συμβιβασμό και δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω το έργο των εισηγητών όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ορισμοί που προβλέπονται πρόκειται να απαγορεύσουν κάποια εντομοκτώνα τα οποία χρησιμοποιούνται και είναι πολύ σημαντικά για τη γεωργία. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν αρκετέ τέτοιε ενεργέ ουσίε Γεωργίου, τόσο ώστε να μπορούν να καταπολεμήσουν οποιαδήποτε ασθένεια πλήση την παραγωγή. Η παραγωγή, συγγνώμη, το, το, το πρόβλημα δεν είναι το προϊόν, το πρόβλημα είναι η κακή του χρήση. Η Ισπανική συνιστόσα του ΕΛΚ υποστηρίζει την πρόταση για έκθεση αξιολόγησης και συμφωνούμε με την τροπολογία που λέει ότι θα πρέπει κάποια ε, προϊόντα τα οποία βοηθούν ιδιαίτερως να μην απαγορευτούν. Θα πρέπει επομένω να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μείωση της παραγωγής διατροφικών προϊόντων και θα πρέπει να ε, υπάρξει αυστηρή ρύθμιση των εισαγών για κάποια προϊόντα τα οποία εμείς δεν παράγουμε. Robert Sturdy. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω μόνο για την έκθεση Μπράιερ και επ' αυτής να πω στην Κομισιόν γιατί είστε κατά μιας έκθεσης αξιολόγησης. Τι σας ανησυχεί τόσο πολύ και δεν θέλετε να γίνει έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις επιστημονικές που να καταδεικνύουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι επικίνδυνα για την υγεία. Κάποια προϊόντα είναι, αλλά εσείς πόρευσατε ένα σωρό προϊόντα απογορεύεται κάποια προϊόντα που δεν είναι επικίνδυνα. Και το τριαζόλ. Αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα σιτήρα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτύχατε σε αυτό το σημείο, το λέω και το εννοώ. Αποτύχατε και ξεπουλήσατε τον κόσμο όσον αφορά το να σταματήσετε τις εισαγωγές των μεταλλαγμένων. Και το έχετε παραδεχθεί αυτό. Επίσης αποτύχατε σε σχέση με τη δική μου έκθεση όσον αφορά τα τα, τα, τα ανώτατα επίπεδα των καταλήπων. Θα ήθελα να μου πει και η παρακαθημένη σας ότι τι πιστεύει, αλλά δεν ακούει γιατί μιλάει. Τι έγινε με αυτά τα ευρήματα στα σούπερ μάρκετ όσον αφορά αυτά τα κατάλοιπα. Καλά, θα απαγορεύσετε τη δική μας παραγωγή. Για τις αγωγές όμως τι λέτε, λέτε δεν πειράζει έτσι κι αλλιώς θα μπουν αυτά τα προϊόντα, οπότε ας μην κάνουμε τίποτα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όμως η γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πιο υπεύθυνοι που υπάρχουν σε σχέση με την παραγωγή ειδών διατροφής. Με τέτοια νομοθεσία τους βραζιλεύεται, τους υποτιμάται. Κανείς από αυτούς δεν θα χρησιμοποιούσε επικίνδυνα, χημικά επικίνδυνα για την υγεία. Εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι σε δύο χρόνια θα απαγορεύσετε κάτι το οποίο αφορά την παραγωγή των αυγών, των λαβών και αυτά τα κλουβιά λοιπόν θα τα απαγορεύσετε και δεν ξέρω τι θα γίνει θα έπρεπε να δώσετε κάποιο περιθώριο στους παραγωγούς να αποδείξουν ότι είναι υπεύθυνοι και μπορούν να παράγουν ασφαλή προϊόντα ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό στην 25 λέει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Okay. I think perhaps you can start again. Μήπως μπορείτε να ξαναρχίσετε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι η ανεύθυνη χρήση των ζενιοκτώνων. Το πώς θα καταλήξουμε να έχουμε υγιεινή παραγωγή, να μην έχουμε καρκινογόνες ουσίες που να χρησιμοποιούνται, ούτε ουσίες που βλάβουν το περιβάλλον. η Κρίστα Κλάς και η κυρία Μπράιερ συνέταξαν αυτές τις εκθέσεις που είναι ένα θετικό βήμα. Θα πρέπει να γνωρίσουμε το ότι κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια. Γίνονται τώρα καινούργια βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος των γεωργών, των καταναλωτών. Έχουμε κάποιους στόχους συγκεκριμένους. Έχουμε Επίσης, αυτές οι διατάξεις που αφορούν αυτή την κοινοποίηση προς τους γειτονιάζοντες γεωργούς που έχει σημασία για τη μελισσοκομεία. Πάντως, θα μπορούσαμε να επιφέρουμε ακόμη περισσότερες βελτιώσεις στην νομοθεσία να μην χρησιμοποιείται επομένω χημικά και να υπάρχει βιολογική γεωργία. Πάρε δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, επιτροπή. Να σας πω λιγότερο από ένα χρόνο πριν ε, συζητούσαμε εδώ τι θα κάνουμε για την ε, παγκόσμια ασφάλεια σε τρόφιμα και αν υπήρχαν αρκετά τρόφιμα στον κόσμο και μας ανησυχούσε τρομερά και φοβερά. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά συζητάμε αυτή την ονομοθεσία σήμερα που έχει τι πιθανότητε να περιορίσει την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και ένα ηθικό δίδαγμα για την παραγωγή τροφίμων, γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν εμεί εδώ στην Ευρώπη δεν παράγουμε φαγητό, ε, μάλλον μπορούμε να πληρώσουμε γι' αυτό, αλλά ο αναπτυσσόμενος κόσμος όχι. Όχι μόνο τα δημητριακά αλλά και οι πατάτες υποφέρουν από αυτά ε, τα παράσιτα. Ήταν δύο από τα χειρότερα καλοκαίρια που έχουμε δει ποτέ στην Βόρεια Ευρώπη. Χρειάζεται το τριαζόλι για να περιορίσουμε τα παράσιτα και αν ο κόσμος στην Ευρώπη δεν φάει πατάτες, τι θα φάει. Ρύζι, Επίτροπε. Ρύζι και ζυμαρικά. Και σίγουρα το ρύζι είναι αυτό το οποίο λείπει από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επιπλέον αυτό που είπε ο κύριος Στέρντι, πολλά από αυτά τα ζανιοκτώνα ή μικητοκτώνα, αν δεν χρησιμοποιηθούν καλά, σωστά και αν χρησιμοποιηθούν σωστά, παράγουν πολύ καλά τρόφιμα τώρα εσείς μου λέτε ότι θα σταματήσετε τις εισαγωγές τροφίμων και ότι εκεί δεν θα τα ψεκάζουμε αυτού του είδους τα χημικά, μα δεν τα καταφέρατε γιατί μπορείτε να δοκιμάσετε τα δημητριακά σας όσο θέλετε όταν έρχονται από το λιμάνι του Ρότερνταμ, αλλά εκεί δεν θα βρείτε κανένα κατάλοιπο. Πραγματικά θα πρέπει να ξυπνήσουμε και να πούμε ότι εμεί στην Ευρώπη πρέπει να φτιάξουμε τρόφιμα, παράγουμε τρόφιμα και με ασφαλή τρόπο. Να διασφαλίσουμε τον την μείωση των χημικών που χρησιμοποιούμε, αυτό το κάνουμε ήδη, και επίση να, το... να το κάνουμε με τρόπο ώστε οι Γεωργοί να μάθουν να αναψεκάζουν σωστά Πράγμα που επίσης κάνουμε. Παρακαλώ λοιπόν κάντε μια σωστή εκτίμηση, ε, αξιολόγηση μάλλον επιπτώσεων. Είχαμε τα δύο χειρότερα καλοκαίρια που έχουν ποτέ καταγραφεί και πραγματικά ε, σας εκλυπαρώ να κάνετε μια σωστή αξιολόγηση επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Επί του κανονισμού, παρακαλώ. Ο κύριος Στίβαν μου πρόσφερε τα δύο του λεπτά και μια που αποξιάζει μπορώ να τα πάρω. Πρόεδρε. Παρακαλώ. Σα mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι υπερβολικές απαιτήσει, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπη, καθίστησαν δύσκολο να δούμε ποιο είναι η γεγονό και τι είναι παραμύθι στην διάρκεια της συζήτησης αυτής. Πράγματι χρειάζεται ανάγκη ελέγχου της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Το δεχόμαστε όλοι. Και αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνα και για τον χρήστη και για το περιβάλλον. Αν χρησιμοποιηθούν όμως φορά και έχουμε το ανώτατο όριο καταλήπων, ο ε, κίνδυνος είναι ελάχιστος και για τον κανονιτή είναι ανύπαρκτος. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ποιε είναι ουσιαστικέ ε, ουσιαστικά, ε, ε, ουσιαστικές ιδιότητες συγγνώμη, των ουσιών αυτών. Εκεί θα πρέπει να βασιστούμε. Το ενόπνευμα, παραδείγματο χάρη. Το, το καθαρό ενόπνευμα είναι επικίνδυνο. Αν πιει κανένα καθαρό ενόπνευμα, ξέρει τι γίνεται. Άμα όμω το διαλύσουμε σε 4%, 12% και σωστά χρησιμοποιούμε, έχει ένα ελάχιστο κίνδυνο. Δύο διαφορετικά θέματα. ο επιστημονικός ε, ο ορισμός έχει ήδη αναφερθεί για, τους, ε, για τις ε, ουσίες που έχουν επιπτώσεις ενδοκρινώς. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να αναπτυχθούν καινούρια προϊόντα. Εγώ θα καλέσω την σχετική βιομηχανία να εξετάσει τον τομέα, να επενδύσει τον τομέα αυτό. Και βέβαια όσον αφορά την, το να επιτρέψουμε την εισαγωγή των προϊόντων αυτών που παράγονται με τα ε, φυτοφάρμακα που απογορεύουμε στους γεωργούς μας δεν είναι σωστό. Γιατί αυτό δεν είναι ισορροπημένο. Η λύση έχει βελτιωθεί, αλλά εξακολουθεί να μην είναι ισορροπημένη, αλλά θα μπορούσα ίσως να τη δεχτώ. Ευχαριστώ. Πρώτα σε ευχαριστώ. Περνάμε στο Catch the Eye. Ένα λεπτό. Κονμπέργκ. Ευχαριστώ i wish to highlight the importance of explaining to affected stakeholders early on in the legislative process the reasons why it is necessary to regulate. Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο χρειάζεται τέτοια νομοθεσία και εγώ άκουσα κάποιους ε, οι οποίοι ε, ανήκουν στον κλάδο στην εκλογική μου περιφέρεια διότι ο κόσμος πιστεύει ότι αυθαιρετούν οι Βρυξέλλες και από τα πάνω επιβάλλονται κάποια, κάποιες ρυθμίσεις. Θα έπρεπε περισσότερο να εξηγούμε σε όλους τους εμπλεκόμενους και να μην τους κατηγορούμε και έτσι να εμφανιζόμαστε ως οι γραφειοκράτες των Βρυξελών. Τα κράτη-μέλη μπορούν πάνω σε αυτό να κάνουν κάτι, μπορούν να εξηγήσουν το τι ισχύει στα κράτη-μέλη, έχουν τους κατάλληλους πόρους, που είναι σημαντικό γιατί Εκείνοι παράγουν το φαγητό το οποίο τρώμε, να μην βάζουν φραγμούς δραστηριότητας από υπερβολική νομοθεσία. Θα πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να είναι πιο ισόρροπη, να λαμβάνει υπόψη τα πάντα. Το περιβάλλον και τα συμφέροντα των καλλιεργητών και τους καταναλωτές. Όλους λοιπόν αυτούς να τους λάβουν υπόψη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει συνάδελφος Σουζάννα Ρόιτοβα. Παρακαλώ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 Ε, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη για το γεγονό ότι είναι ο καθήκον μα να, προς τους καταναλωτές να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη χρήση των ε, φυτογενομικών, τοξικών προϊόντων στα φυτογενομικά προϊόντα. Ωστόσο, γνωρίζω <coughs> ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ώστε να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη καλύτερων παρασιτοκτόνων και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε εξαιρέσεις για κάποιες χώρες και ορισμένες χώρε άλλε θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό και επιμένω τα κράτη κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει χωρίς συμβιβασμούς να ελέγξουν τι συμβαίνει και τα εισαγόμενα προϊόντα ε, δεν, ε, θα, δεν ελέγχονται. Ακόμα και τα λουλούδια θα πρέπει να ελέγχονται ε, αυτά που εισάγονται. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τον στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης, να συμφωνήσω με αυτούς που επικρίνουν, που λένε ότι επειδή δεν έκανε η Κομισιόν αντίκτυπο, μελέτη αντικτύπου, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το, σε επιπτώσει αυτής της νομοθεσίας. Ο κύριος Μπάτον. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει κάνει εξαιρετική ζημιά στη Βρετανική Γεωργία και τεράστιο κόστος οικονομικό. Και τώρα έχουμε αυτή την πρόταση για τη παρασιτοκτόνα. Εκτιμάται ότι αυτή η οδηγία μπορεί να σημαίνει την κατάργηση 15% των παρασιτοκτόνων. Αυτό θα περιορίσει τις εσοδιές από, 28 έως 86%, η πατάτα 23 μέχρι 56% και ορισμένες άλλες οδιές από 25 μέχρι και 75% θα μειωθούν. Αυτό θα έχει ως επιπτώσεις ε, να, ε, να ανεβούν στα ύψη οι τιμές λιανικής τιμής και ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να πληρώσει το τρόφιμα. Εγώ διερωτώ με αν οι συγκητές μπορούν να μας πούν τα ονόματα, την ταυτότητα, έστω και ενός ανθρώπου που έχει... Ε, ε, ζημιωθεί ή έχει πεθάνει λόγω των επιπτώσεων αυτών των ε, που Εγώ μπορώ να σας πω πολλούς από τους κατοίκους της περιφερειάς μου που δεν μπορούν πια να πληρώνουν ε, τα φρούτα τους. Ευχαριστώ. Πείτε η χρησιμοποίηση αυτών των φυτογενομικών προϊόντων είναι το αντικείμενο αυτής της οδηγίας και θα πρέπει να χαιρετήσουμε το ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και τα κράτη-μέλη. Έχουμε θέσει τις προστατευτικές περιοχές, συμφωνώ, αλλά επίσης συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια προγράμματα εθνικά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει το περιθώριο εφαρμογής των εθνικών διατάξεων. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο το ότι έχουμε και συμβασμό και για τους ψεκασμούς από αέρος όμως είναι εύστοχη αυτή η ρύθμιση που αφορά την απαγορεύση των ουσιών των επικινδύνων για την ανθρώπινη υγεία όμως ε, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά το τι γίνεται με τις τρίτες χώρες και πώς θα έχουμε την δική τους χρήση χημικών είναι σωστό, τον έχουμε δει αυτή την έγκριση και την ε, αδειοδότηση. Ε, δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικό για να καταλάβει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα ε, η Ουγγαρία αποτελεί ενιαία ε, ζώνη, υπάρχουν και τα προβλήματα της Ιλλανδίας. Πρόεδρος, δίνει το λόγο στον επόμενο. Ρένα Τράκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα θέμα το οποίο δεν εθίγει σήμερα εδώ. Με τελευταία αναλύση θα έχουμε πάλι πετύχει, ελπίζω, ένα λογικό συμβασμό στην Ευρώπη. Αλλά τι κάναμε καθοδόν. Ας θυμηθούμε ε, τις ε, μακρόχρονες συζητήσει με κατηγορίες από πλευράς και από τις άλλες και από την άλλη. Όλα αυτά βέβαια πέρασαν με ενθουσιασμό στα ΜΜΕ και τα ΜΜΕ έτσι οδήγησαν σε ανασφάλεια τους καταναλωτές, ε, όλοι μπορούσαν να συμφωνήσουν, δεν τα ε, κάνει σωστά αυτά που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εις βάρος των ε, πολιτών, δεν είναι υπέρ των πολιτών. Τώρα πετυχαίνουμε ένα συμβιβασμό στο οποίο θα υπάρχει ευρεία συνένεση. Τι θα κάνουμε τελικά όμως, τι θα έχουμε στα χέρια μας για το καναλτή, τίποτα σχεδόν. Σικιέρσκι, πρόεδρος. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συζητούν ζητήματα που αφορούν την διατροφική ασφάλεια. Είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε σαφήνεια των ρυθμίσεων. Να είναι κατανοητά αυτά τα νομοθετήματα να βασίζονται σε κάποια επιστημονική γνώση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα η αγροτική παραγωγή. Θα πρέπει επομένω να υπάρξει κάποιο είδους παρακολούθηση του τι αποτελέσματα θα φέρει αυτή η νομοθεσία. Θέλουμε να υπάρχουν επιστημονικά θεμέλια για αυτές τις ε, ρυθμίσεις και έτσι να έχουμε εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα προϊόντα προστασία είπαμε της δημόσιας υγείας αλλά να μην αυξηθούν ε, οι δαπάνες της παραγωγής. Μήπως τώρα θα επιβαρυνθεί και η κοινή αγροτική πολιτική όσον αφορά την οικονομική πλευρά του θέματος. Έχουμε και επιστροπολογίες και θα τις υποστηρίξουμε, είναι δικές μου και άλλων συναδέλφων. Νίκολσον. Πρόεδρε, προβληματίζομαι βαθιά όσον αφορά αυτό το νομοθέτημα να γραφεί στα πρακτικά του συμφωνώ με τις τροπολογίες στέλνει, τις προσυπέγραψα και θα τις επιψηφίσω. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν κάπως τον κλάδο. Βεβαίως και χρειάζεται τέτοια νομοθεσία. Θα πρέπει όμως να είναι εύστοχες οι ρυθμίσεις για να μην παραβλάψουμε την παραγωγή. Χρειάζεται και μια καλή έκθεση για τις επιπτώσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία πάνω στα οποία να στηριχτούμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εισαγωγές. Έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά η Κομισιόν. Άλλα επιβάλλει στο εσωτερικό και άλλα επιτρέπει για αυτούς οι οποίοι φέρουν προϊόντα από το εξωτερικό. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Πετάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Επίτροπος κ. Δήμας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλους εκείνους οι οποίοι πήραν ε, το λόγο απόψε στη σημερινή συζήτηση ε, και ιδιαίτερα για τις πολύ επικοδομητικές τους παρεμβάσεις. Με βάση το κείμενο που συμφωνήθηκε και το οποίο είναι συμβιβασμός και μάλιστα πολύ επιτυχημένος, τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται να καταρτήσουν εθνικά σχέδια δράσης στα οποία θα καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι για τον περιορισμό των κινδύνων με τα εθνικά σχέδια δράσης τα κράτη μέλη θα οφείλουν επίσης να παρακολουθούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων που έχουν κατά ε, προκαλέσει συγκεκριμένα προβλήματα και να καθορίζουν στόχους μείωσης της χρήσης ορισμένων από αυτά. Ε, πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου ε, και το οποίο θα έχει πέραν των, προστασία της προστασίας της των Ευρωπαίων πολιτών ε, και του περιβάλλοντος και οικονομικά ωφέλη από το ότι λιγότερη θα είναι η δαπάνη ε, για την ε, υγεία και στα εθνικά συστήματα υγείας καθώς επίσης, καθώς επίσης και από τη μικρότερη χρήση των φυτοφαρμάκων που θα προκύψει από την παρούσα νομοθεσία. Εκτός από τα εθνικά σχέδια δράσης η προτινόμενη συμβιβαστική δέσμη περιέχει και ορισμένες άλλες σημαντικές ε, πτυχές. πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης. στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών δίδεται προτεραιότητα σε άλλες μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας. ενισχύεται η προστασία των περιοίκων και των διερχομένων προσώπων. πιο συγκεκριμένα τα εθνικά σχέδια δράσης θα μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση των ατόμων που μπορεί να εκτεθούν σε μετακινούμενο νέφος που δημιουργείται από τους ψεκασμούς ενώ οι εκτάσεις που πρόκειται να ψεκαστούν από αέρος δεν θα πρέπει να γυτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. όλοι οι διανομής φυτοφαρμάκων και όχι μόνο όσοι πολλούν σε επαγγελματίες χρήστες θα μεριμνούν ώστε κάποια άτομα από το προσωπικό τους να διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό επάρκειας που βεβαίως ε, επειδή έγινε μια παρατήρηση σχετικά ε, θα είναι αμοιβαία αναγνωρίσιμο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα φυτοφάρμακα και να είναι στη διάθεση των πελατών για παροχή συμβουλών. Από την υποχρέωση αυτή θα απαλλάσσονται μόνο ορισμένες κατηγορίες μικροδιανομέων. Σε ό,τι αφορά στην απογόρευση του αεροψεκασμού βρέθηκε συμβιβαστική λύση για τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων εξαίρεσης. Η εξαίρεση θα ακολουθεί διαδικασία που θα περιλαμβάνει δύο βαθμίδες. Πρώτα, την κατάρτιση γενικού σχεδίου αεροψεκασμού, το οποίο θα υπόκειται σε ρητή έγκριση των αρχών και στη συνέχεια την υποβολή ειδικών αιτήσεων αεροψεκασμού κατά περίπτωση οι οποίες θα υπόκεινται στις προϋποθέσεις έγκρισης του γενικού σχεδίου κλείνοντας ε, κυρία πρόεδρε η επιτροπή είναι ικανοποιημένη από την έκβαση των διαπραγματεύσεων και για το λόγο αυτό είναι σε θέση να αποδεχθεί πλήρως τις προτινόμενε συμβιβαστικές τροπολογίες. σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για την καρποφόρα συμμετοχή σας σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Κομισιόν έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το φάκελο και εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για το υψηλότερο επίπεδο δημόσιας υγείας που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Έχουν γίνει μακρές και δύσκολες συζητήσεις κατά τη διάρκεια του τριμερούς ε, διαλόγου, που, τις οποίες ε, με μεγάλη προσήλωση και δεξιο, επιδεξιότητα χειρίστηκε η εισηγήτρια και την ευχαριστώ γι' αυτό. Η Κομισιόν υποστήριξε την κοινή θέση και μπορεί τώρα να υποστήριξει την πρόταση, καθώ αυτή προκύπτει από τη δεύτερη ανάγνωση. Όλε οι καινοτόμε πτυχέ τη πρόταση έχουν διατηρηθεί ιδιαίτερα το κριτήριο έγκρισης που θα διασφαλίσει ότι επικίνδυνες ουσίες που δημιουργούν ψηλό κίνδυνο για τη δημόσια θα καταργηθούν ή θα αντικατασταθούν με ασφαλέστερες εναλλακτικέ λύσεις ε, βελτιωμένη αμοιβαία αναγνώριση και υποκατάσταση ορισμένων προϊόντων από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Αλλά δεν ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν Σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν, μόνο το 4% των ουσιών που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά θα εξαφανιστούν επειδή ε, αποτελούν ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες και μόνο το 2% διότι είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή. Το σύνολο των ε, ενεργών ουσιών που αυτή τη στιγμή δηλαδή βρίσκονται στην αγορά, κυκλοφορούν στην αγορά και που θα πιθανότατα δεν θα εγκριθούν από τον νέο κανονισμό αναμένεται να είναι χαμηλότερο των 25. Αυτή η αξιολόγηση έχει επιβεβαιωθεί από την έκθεση της Σουηδικής ε, Υπηρεσίας Χημικών και είναι και σύμφωνη με την αναθεωρημένη αξιολόγηση κινδύνου από την ε, Βρετανική Διεύθυνση Ασφάλειας ε, Παρασυτοκτόνων. Επιπλέον να τονίσω ότι νέα κριτήρια θα ισχύσουν για τις ήδη κεκριμένες ουσίες μόνο με την ανανέωση της ε, αδειοδότησής τους και ε, οι περισσότερες από αυτές θα αναθεωρηθούν μόνο το 2016. Άρα λοιπόν η βιομηχανία θα έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να ανακαλύψει και να αναπτύξει νέες και ασφαλέστερες ουσίες. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια που έγιναν σε σχέση με τα εισαγόμενα τρόφιμα. Να σας θυμίσω ότι από το 2008 έχουμε τον κανονισμό για τα μέγιστα επίπεδα καταλήπων που ισχύει πλήρως, που έχει τεθεί πλήρως εφαρμογή. Ακόμα δηλαδή και αν μια ουσία δεν είναι εγκεκριμένη για τη χρήση σε προϊόντα φυτοπροστασίας στην Ένωση, τα με επίπεδα καταλήπων για αυτές τις ουσίες ορίζονται σε το επίπεδο της ανείχνευσής τους. Αυτά τα MRL ισχύουν για την ε, κοινωτική παραγωγή αλλά και για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ζωοτροφές. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μια ενεργή ουσία δεν μπορεί να εγκριθεί στην Ένωση και για τον πιθανό κίνδυνο στους καταναλωτές. Μία από αυτές τις αιτίε είναι ο κίνδυνος καταναλωτές. Άλλες μπορεί να συνδέονται με περιβαλλοντικά ζητήματα ή την προστασία των εργασομένων που είναι θέματα τα οποία επιπτούν στην ε, κυριαρχία των χωρών όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα ζυζανιοκτώνα, η παραστοκτώνα. Σε αυτές τις περιστάσεις η χρήση των παραστοκτώνων τα ζυζανιοκτωνα οι παραστοκτωνα σε αυτες τις περιστασεις η χρηση των παραστοκτωνων μπορει να μην είναι αποδεκτή για εμά, αλλά οι σοδιές που έχουν υποστεί κατεργασία και που δεν που μπορεί να μην παρουσιάζουν απαραίτητο κίνδυνο για τους ε, καταναλωτές. Γι' αυτό και μια τρίτη χώρα που θέλει να εξάγει τέτοιου είδους κατεργασμένες ουσίες στην Ένωση μπορεί να ζητήσει για μια ανοχή στις εισαγωγές από τη στιγμή που μπορεί να υποβάλει στοιχεία που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση αυτών των αγαθών και ότι αυτά τα στοιχεία θα αξιολογηθούν θετικά από την ΕΦΣΑ και θα υιοθετηθούν επισήμως από την κοινοτική νομοθεσία. <laughs> Αυτή είναι η θέση, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τα εισαγόμενα αγαθά. Τώρα, αν επανέλθουμε στην οδηγία την οποία προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε. Η Κομισιόν θεωρεί πως η τελική συμβαστική λύση είναι ισορροπημένη, πως επιτυγχάνει τους στόχους της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και ε, διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των παραστοχτών για τους ε, γεωργούς. Ε, αυτή τη στιγμή προσβλέπουμε στην τυποποίηση είναι ε, ολοκλήρωση μάλλον τη συμφωνία Δεύτερη Ανάγνωση, που είναι βεβαίω ένα πολύ καλό τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με προοπτική για του πολίτε μα, καθώ αυτό ωφελεί την υγεία του. Είναι επίση ε, περιστεύουμε, επόφελε για του γεωργού μα γιατί διασφαλίζει την παραγωγή του μέσω συγκεκριμένων μέτρων όπω η προώθηση των ασφαλέστερων προϊόντων. Αυτό που επετεύχθη είναι πολύ σημαντικό. Επετεύχθη από όλους μας μαζί και και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η διοργανική συνεργασία μπορεί άμεσα να ωφελήσει τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία μου, θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Κλάσσα. δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα με σύγχρονη λυτική μπορούμε να βρούμε ε, ένα κουτάλι ζάχαρης μέσα σε μια τεράστια λίμνη. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Πώς θα τις εκμεταλλευτούμε. Χρειαζόμαστε νομίζω αντικειμενικά στοιχεία ε, κινδύνου που θα ισορροπούν τις ε, δικαιολογημένες απαιτήσει για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και επίσης την προστασία της επιστημονικής, ε, επιστημιστικής συγγνώμη, ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα αυτό ετέχθη. Δεν νομίζω ότι εδώ θα απέρκες απαιτήσεις από την Κομισιόν. Δεν χρειάζεται να μας πείτε ότι δεν απαγορεύονται δύο ουσίες ή τέσσερις ουσίες σε αυτό το μέσο στο άλλο τομέα, στο σύνολο 25. Όχι, χρειαζόμαστε σημαντικά ε, στοιχεία για το πώς πληρούνται όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τα επιστημονικά κτίρια και νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει τώρα να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της νέας αυτής νομοθεσίας σωστά για να ξέρουμε ποιες είναι τελικά οι επιπτώσεις. Και θα πρέπει να το συνοδεύσουμε αυτό γιατί τα επιστημονικά αποτελέσματα δεν είναι στάσιμα, εξελίσσονται. Ο συμβιβασμός δίνει πολλά στοιχεία για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα φάρμακα. Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και απαιτεί από τα κράτη-μέλη ε, συγκεκριμένα μέτρα για την εξασφάλιση αεφόρου χρήση των φυτοφαρμάκων. Ω εισηγήτρια θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Καταφέραμε διαφορετικές ε, θέσεις εκκίνησης να τις συμβιβάσουμε και να πετύχουμε αυτόν τον συμβιβασμό. Στο ε, νέο έτος ελπίζω να έχουμε πιο θετική σκέψη. Γιατί αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι τα φυτοφάρμακα μας εξασφαλίζουν επαρκή και υγιή τρόφιμα και υγιές περιβάλλον. Ευχαριστώ. Πρώτα, σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπράιερ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έντονη συζήτηση. Δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι κατά γνώμη μου εξακολουθούμε να έχουμε εδώ ένα ε, ορόσημο για την πολιτική της Ευρώπης γιατί τώρα η Ευρώπη είναι εκείνη που ξεπερνάει που είναι ο ηγέτης σε διεθνές επίπεδο που μας κάνει να εγκαταλείψουμε αυτά τα πολύ επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό στον κόσμο και μπορεί να είναι περήφανη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όσον αφορά τα διάφορα επιχειρήματα που ακούσαμε ότι δεν έχει επιληθεί το θέμα των εισαγωγών. Δεν είναι σωστό αυτό. Έχει λυθεί το πρόβλημα των εισαγωγών. Γιατί με την απαγόρευση των, ε, των ε, ουσιών αυτών, ε, αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες είναι παράνομες. Εάν εισάγουμε πολικευτικά ή ανθή θα πρέπει αυτά να τηρούν τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν μέσα στα πλαίσια του κανονισμού για τα ελάχιστα κατάλοιπα, για τα μέγιστα συγγνώμη κατάλοιπα, βρεθούν κάποιες ουσίες, αυτά τα τρόφιμα είναι παράνομα. Αν πούμε οι μπανάνες από την Κωνσταντίνα περιλαμβάνουν κάποιες ουσίες που σε εμά είναι απαγορευμένες, είναι παράνομη κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έχουμε μια καλή λύση γιατί Χρησιμοποιούμε όχι μόνο αυτούς τους κανονισμούς εδώ, αλλά και τους κανονισμούς για τα μέγιστα κατάλοιπα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Η Επίτροπος μάλιστα έχει την καλοσύνη να το αναφέρει. Αν σκεφτούμε ότι στην πρώτη μελέτη του ΠΕΣΤΕ έλεγε ότι θα πρέπει το 80% των φυτοφαρμάκων να εξαφανιστούν από την αγορά. Τώρα όμως μειώσαμε σημαντικά τον αριθμό αυτό δυστυχώς δεν αφαιρθήκατε καθόλου στην αναβελτίωση αυτή της μελέτης πέσα. Λοιπόν, Σάπαρ, παρακαλώ, για να τελειώσει πια αυτή η κινδυνολογία. Ας δεχτούμε αυτόν τον συμβασμό που είναι προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Διακόπτη, Πρόεδρος. Κυρία Μακίνες, διαδικαστικό. Μάλιστα, έχω ένα διαφορετικό γιατί νομίζω ότι πολλοί ακούν, ε, μιλάνε και δεν ακούν. Άκουσα τι είπε η, η Επίτροπος για τις αγωγές και τι είπε και η συγγήτρια για τις αγωγές. Είπαμε, οι παραγωγοί στην Ευρώπη θα απαγορευτεί να χρησιμοποιούν κάποιες ουσίες. Οι ξαδέλφοι τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τις χρησιμοποιούν. Στα τρόφιμα δεν υπάρχει κανένα λοιπόν όμως συζητάμε για ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τους παραγωγούς της Ευρώπης. Ίσως κάποια άλλη στιγμή να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και όχι αυτά τα ασαφή στα οποία κινούμεθα αυτή τη στιγμή. La discussion commune Bon, nous allons pas recommencer. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Προφανώς είναι αυτό. Δεν θα πρόκειται να αρχίσουμε από το μηδέν πάλι. Κυρία Μπράγερ, 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εξήγησα και η Επίτροπος εξήγησε ξεκάθαρα. Αν δεν ακούτε ή αν δεν θέλετε να ακούσετε ότι λύσαμε το πρόβλημα, γιατί δεν είναι σύμφωνο με τη δική σας εκστρατεία κατά του κανονισμού. Ε, τι να κάνω. Δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα, αλλά μπορώ να ξαναπώ ότι είναι ασφαλές διότι έχουμε τον κανονισμό για τα μέγιστα επίπεδα καταλήπων. Έχει λυθεί λοιπόν το πρόβλημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί κανένας να εμπορευτεί μία ουσία που δεν επιτρέπεται να εμπορευτεί. Τελεία. Bien, nous allons pas recommencer le débat. Je vous engage. Λοιπόν, λέει πρόεδρος, αν θέλετε να συνεχίσετε τη συζήτηση, στο διάδρομο παρακαλώ. Έκλεισε η κοινή συζήτηση εδώ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Τώρα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, θα περάσουμε στην προεκλογική ερώτηση προ την Κομισιόν για το σχέδιο δράση για την κινητικότητα. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο καταρχήν στον συντάξαντα, τον κύριο Κώστα, για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή της οποίας εσείς είστε μέλος επανειλημμένως ανακοίνωσε το πρόγραμμά της για την αστική κινητικότητα και το οποίο θα έπρεπε να υποβληθεί από τον περασμένο φθινόπωρο στην Κοινοβούλιο